Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας. Please be seated. If you're all ready. Αν είσαστε όλοι έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και τώρα συνεχίζω στα ισπανικά, λέει ο πρόεδρος. Σας χαιρετίζω όλους. Καλώς ήρθατε. Προς όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές, κυρίους και κυρίες, από την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη, τη ΛΥΜΠΕ, των νομικών υποθέσεων, τη Γιούρη δηλαδή. Και ε, καλωσορίζω και στους ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Καλώς ήρθατε όλοι, κυρίες και κύριοι. Και καλώς ήρθατε και εσείς, κυρία Ρέντιν. Που είναι η προτινόμενη Επίτροπος για ένα χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικό όσον αφορά τη δομή της νέας Επιτροπής. Πρόκειται για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Σήμερα είμαστε εδώ τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές λοιπόν, αναφέρθηκα σε αυτές. Η ακρόαση θα κρατήσει τρεις ώρες. θα ξεκινήσουν οι πρόεδροι των ε, Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, εγώ ίδιος, και της Επιτροπής Γιούρη. Ο κύριος Λένε δηλαδή και η πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών, η κυρία Σβένσον. Όμως, έχουμε φροντίσει για μια διάρθρωση έτσι ώστε μία ώρα και ένα τέταρτο θα εξετάσουμε, την πρώτη ώρα δηλαδή και ένα τέταρτο, θα εξετάσουμε την προτινόμενη Επίτροπο για τα θέματα δικαιοσύνης στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σύμφωνα με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων θα έχουμε μία ώρα ερωτήσεων και απαντήσεων με 20 ερωτήσεις. Μία ώρα και ένα τέταρτο θα κρατήσει αυτό το κομμάτι όπως σας είπα και πριν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα αναγκαστώ πολύ αυστηρός με το χρόνο. Θα φροντίσω πολύ αυστηρά να τηρηθεί ο χρόνος. Ένα λεπτό για την κάθε μία από τις 20 ερωτήσεις και δύο λεπτά για την απάντηση της κάθε ερώτησης. Οι ευρωβουλευτές που θα πάρουν το λόγο πρέπει να το ξέρουν αυτό. Εκπροσωπούν τις πολιτικές ομάδες σύμφωνα με το σύστημα DONT. Με τη σειρά θα πάρουν το λόγο Υπάρχει σειρά ήδη και όπως σας είπα και πριν να φροντίσετε να τηρήσετε το χρόνο σας. Ένα λεπτό ο καθένας. Μετά το σφυράκι μου θα χτυπάω και η κυρία Ρέντινγκ παρακαλώ επίσης να τηρήσει το χρόνο δύο λεπτά απάντηση στην κάθε ερώτηση που θα ακούσει. Ξέρω ότι οι εργασίες μας είναι πολύ ενδιαφέρουσες, περιλαμβάνουν πάρα πολλά θέματα. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ της Λισαβόνας περνάει σε νέα φάση, κυρίως στα θέματα δικαιοσύνης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως επίσης και η ισχύ του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλάζει επίσης κάπως το σκηνικό. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω πρώτα από την κυρία Ρέντινγκ να πάρει το λόγο για 10 λεπτά για να κάνει μια αρχική παρουσίαση και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ κυρία Ρέντινγκ. Αγαπητά μέλη, είναι η τρίτη φορά που έχω την τιμή να είμαι εδώ μπροστά σας σαν υποψηφία επίτροπος. Οι ακροάσεις για μένα είναι μια πολύ ισχυρή στιγμή της δημοκρατίας. Εδώ δείχνουμε ότι είμαστε πράγματι υπόλογοι, δείχνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι για συζήτηση και δείχνουμε στους πολίτες μας ότι έχουμε εδώ μια μορφή δημοκρατίας μοναδική δεν υπάρχουν πολλά κοινοβούλια στον κόσμο τα οποία έχουν καταφέρει να κερδίσουν τη μάχη αυτή και να αποκτήσουν το δικαίωμα να θέτουν ερωτήσεις προς τα μέλη της κυβέρνησής τους. Έχουμε δώσει μάχες γι' αυτό και εγώ σαν βουλευτής έχω δώσει μάχες σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Και είμαι θύμα σε εισαγωγικά αυτής της διαδικασίας σήμερα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και υπερήφανη για αυτήν την πολύ σχηρή στιγμή της δημοκρατίας. Και για πρώτη φορά παρουσιάζουμε μπροστά σας σαν η πρώτη επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και θέματα που αφορούν τον πολίτη και την ιδιότητα του πολίτη. Σε, ορισμένες, λοιπόν, σε ορισμένα επίπεδα και του Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει γύρω από αυτές τις μορφές επικοινωνίας. Έχουν απογοητευτεί στο παρελθόν. Οι προσδοκίες τους δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί ποτέ δεν υπήρχε και πολιτική βούληση αλλά κυρίως δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα πολιτικά μέσα. Ενθυμούμε όταν ήμουν αντιπρόεδρος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Νομικών Υποθέσεων δεν έφταναν ποτέ σε εμάς, ελαμβάνοντο πίσω από πόρτες ερμητικά κλειστές. Δεν υπήρχε διαφάνεια εκείνη την εποχή το Κοινοβούλιο δεν είχε σχεδόν τίποτα να προσθέσει στα θέματα που άπτονται του λεγόμενου τρίτου πυλώνα. Και οι ευρωβουλευτές ε, είχαν μόνο, θα έλεγα, όνειρα για το τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον. Αλλά από την 1η Δεκεμβρίου ευτυχώς του 2009 τα πράγματα άλλαξαν με τη συνθήκη, τη νέα συνθήκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξει ότι η νέα συνθήκη, η συνθήκη της Λισαβόνας δεν αφορά μόνο τα μεγάλα λόγια αλλά είναι μια ουσιαστικά μια επανάσταση θα έλεγα για τα θέματα, τα εσωτερικά θέματα, τα θέματα της δικαιοσύνης κτλ η συναπόφαση, η διαδικασία συναπόφασης, όπως επίσης και οι νέες διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στο Συμβούλιο με ειδικέ πλειοψηφίες, ε, θα ε, διευκολύνουν πάρα πολύ τον αμοιβαίο σεβασμό των αποφάσεων των δικαστικών ανάμεσα στις διάφορες χώρες και η χάρτα επίσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι στο ίδιο επίπεδο με τη συνθήκη πλέον και αυτό πρέπει να ακολουθηθεί από δράση. Ήταν μακρά η οδός που να φτάσουμε σήμερα εδώ και οι πολίτες δικαιωματικά αναμένουν πλέον από μας να περάσουμε σε δράση και να δώσουμε αποτελέσματα. Είμαι συνεπώς πεπισμένη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας σήμερα σημαίνει ουσιαστικά ένα νέο προσανατολισμό των πολιτικών μας στον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη ή της ηθαγένειας αν θέλετε όχι μόνο σε επίπεδο τυπικό, σε επίπεδο συνθήκης, αλλά σε επίπεδο ουσίας, γιατί η ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη, η ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Είχαμε συγκεντρώσει την προσοχή μας στα θέματα της ασφαλείας κυρίως. Είχαμε, θα έλεγα, ελαφρώς παραμελήσει τη δικαιοσύνη. Η συνθήκη της Λισαβόνας όμως μας δίδει τη δυνατότητα να εξισορροπήσουμε τα δύο αυτά επίπεδα και να φέρουμε στο ίδιο επίπεδο και να συμπεριλάβουμε στην ενασχόλησή μας και τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό το ε, πρότεινε και αναφέρθηκε σε αυτό αναπροσανατολίζοντας την πολιτική ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργώντας και αυτό το χαρτοφυλάκιο που με αφορά σήμερα. εφόσον με επιβεβαιώσετε στα πλαίσια της ανάληψης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, τότε θα βοηθήσω και εγώ έτσι ώστε να αναπροσανατολισθούν οι κοινοτικές πολιτικές στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, προς το συμφέρον του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε από κοινού μαζί με την Σεσίλια Μέλστρομ, την αρμόδια επίτροπο, είναι να καταθέσουμε το πρόγραμμα δράσης για τη Στοχόλμης όπως ονομάζεται θα πρέπει να το ξεκινήσουμε άμεσα. Είναι δύσκολη και μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν άνω των 170 πρωτοβουλειών που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πρωτοβουλίες τις οποίες και εσείς θα εξετάσετε. Συνεπώς έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας ε, για τα επόμενα χρόνια. Πριν περάσουμε στην ουσία των συζητήσεών μας μέσω των ερωτήσεών σας, να μου επιτρέψετε να καταθέσω τρεις κατά προτεραιότητα τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις, α, ε, ε, τις ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας ε, της καθημερινής μας ζωής σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων θα είναι κάτι πολύ υψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων μου και σε σχέση με την καταστολή, την πρόληψη του εγκλήματος και στον τομέα των διεθνών σχέσεων με εταίρους όπως είπα. Δεύτερη προτεραιότητα. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του πολίτη να μετακινείται πραγματικά ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μόνος είτε με την οικογένειά του. Η ελευθερία κίνησης είναι θα έλεγα ο πυρήνας των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην εσωτερική αγορά. Αλλά εδώ είπα τη λέξη αγορά. Εδώ έχουμε μείνει πάρα πολύ στην αγορά και έχουμε ξεχάσει τον πολίτη. Δεν θα πρέπει η έννοια Ευρωπαίος πολίτης να παραμείνει μια αφηρημένη ιδέα, αλλά να γίνει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα για όλους τους πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κοινοτικό νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και αυστηρά. Τρίτον, θα πρέπει επίσης και οι κατηγορούμενοι και οι ύποπτοι για εγκλήματα να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Ξέρετε ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και επίσης έχουμε και τις διαδικασίες τις ανακριτικές της κοινέ, αλλά θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει σχετικά με το δίκαιο των διαδικασιών, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης, με τις συνθήκες φυλάκισης και προσαγωγής και ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του θύματος γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κανένας τομέας της δικαιοσύνης ε, προχωρημένος και καμία αμοιβαία εμπιστοσύνη αν δεν βασιστούμε στις κοινέ αξίες όλοι. Απαιτείται λοιπόν να ενισχύσουμε τα διαδικαστικά στάδια όπως επίσης και τα δικαιώματα των θυμάτων. Εγώ αναφέρθηκα τώρα σε τρία θέματα θα παρατηρήσετε, υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερα όμως και θα επανέλθω σε αυτά κατά τη διάρκεια των ερωτήσεών σας. Thank you. Thank you. Thank you, Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Ρέντινγκ, ε, το λόγο λοιπόν έχει τώρα ο κύριος Μπουζούτιλ ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, ευχόμαι κάθε καλό, επιτυχία στην κυρία Ρέντινγκ και θέλω να πω το εξή. Αν όλα πάνε καλά σήμερα, η κυρία Ρέντινγκ ε, θα είναι για τρίτη φορά επίτροπος, δηλαδή ε, θα έχει ένα σύνολο 15 ετών ως θητεία. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σας ε, ρωτήσω κατά πόσον είσαστε πεπειραμένοι όσον αφορά τις αρμοδιότητες επιτρόπου. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες σας υπάρχει και το θέμα των δικαιωμάτων του πολίτη της ηθαγένειας. Και εμείς ε, προσβλέπουμε στο ότι εσείς ε, θα ενισχύσετε τα δικαιώματα των πολιτών, θα τα καταστήσετε περισσότερο συγκεκριμένα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ζητήσω να μας αναφέρετε τουλάχιστον τρία συγκεκριμένα παραδείγματα, τρία συγκεκριμένα δικαιώματα που προτίθεστε να αποδώσετε στους ε, Ευρωπαίους ε, πολίτες με την ιδιότητά σας της Επιτρόπου. Η κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι διάβασα πολύ προσεκτικά την ε, τόσο σημαντική έκθεση του συναδέλφου σας, ε, κυρίου ε, Λαμασούρ, με τίτλο «Τα δικαιώματα και εφαρμογή των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών». Σε αυτή λοιπόν την έκθεση υπάρχουν τα πάντα. Όλα εκείνα τα κενά, τα οποία πλήττουν τους πολίτες μας όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε πολύ ε, γρήγορα να σας αναφέρω τι θα ακριβώς θα κάνω. Πρώτον, όσον αφορά τον τομέα της ε, δικαιοσύνης. Ε, παράδειγμα, αν είσαστε Φινλανδός που θέλετε να παντρευτεί μία Βρετανίδα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, διότι η Φινλανδία ζητάει ένα πιστοποιητικό που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, έλλειψης εμποδίων κολλημάτων και η Μεγάλη Βρετανία δεν εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό. Άρα δηλαδή για να γίνει αυτός ο γάμος ε, πρέπει το νεαρό ζευγάρι να υπερπηδήσει ένα ε, τεράστιο ε, λαβύρινθο γραφειοκρατικό. Άρα δηλαδή πρέπει να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αναγνώριση των επίσημων εγγράφων και χρειαζόμαστε τα, τα ευρωπαϊκά πρωτότυπα έγγραφα. Ως Επίτροπος, ε, πρέπει να σας πω ότι είχα ε, ξεκινήσει μία πρόταση για την κληρονομιά, για τις κληρονομιές. Ε, για να μπορέσουμε να λύσουμε και το άλλο θέμα, ε, θέλω να σας πω ότι προτιθέμεθα να εκδώσουμε και ένα άλλο έγγραφο ε, που θα εκδοθεί το 2010 και κατόπιν θα ακολουθήσουν νομοθετικής φύσεως ε, πρωτοβουλίες. Εφόσον λοιπόν ήδη αναφέρομαι στα διάφορα έγγραφα και σας ανέφερα και το συγκεκριμένο παράδειγμα των μεικτών γάμων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μεικτοί γάμοι, περίπου είναι οι γάμοι αυτοί ε, και έχουμε περίπου 170.000 διαζύγια σε αιτήσια βάση που σημαίνει περίπου το 20% του συνόλου των διαζυγίων αφορά μικτούς γάμους. Το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο το διαζύγιο, είναι και το θέμα της ε, νομικής ασφάλειας που συνοδεύει το διαζύγιο. Εδώ έχουμε πάρα πολύ θλιβερές ε, ιστορίες και στο Συμβούλιο από το 2006 έχει μπλοκαριστεί η νομοθεσία για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ε, κοιτάξτε, δύο λεπτά έχετε κάθε φορά για να απαντήσετε. Τώρα θα σε επιτρέψετε να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας, αλλά θα ήθελα να σε επισημάνω ότι υπάρχουν ε, αυστηρά κριτήρια όσον αφορά το χρόνο. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Ε, το 2010 θα εκδώσουμε την απαραίτητη νομοθεσία και υπολογίζω στη δική σας τη βοήθεια. Θα προχωρήσουμε με την ε, διπλωματική προστασία και αυτή των προξενείων, έτσι ώστε στο τέλος του 2010 να έχουμε νομικά δεσμευτικούς κανονισμούς. Θα θέσουμε σε ισχύ την οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση που θα προβλέπει, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, και την διαδικασία επί παραβάση. Θα χρησιμοποιήσω αν κρίνθει απαραίτητο και την διαδικασία που προβλέπεται ε, τη σχετική για να ενημερώνονται οι πολίτες. 20 ερωτήσεις θα τεθούν σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων, άρα δηλαδή ε, καταλαβαίνετε ότι ε, υπάρχει περιορισμός χρόνου. Τώρα χρησιμοποιήστε 3,5 λεπτά. Να σας πω λοιπόν, μην το ξανακάνετε, δύο λεπτά στην απάντηση και ένα λεπτό θα έχει στη διαθέσή του κάθε φορά ο ερωτών. Κυρία Ρέντινγκ, κύριος Μωράες, θα είσαστε ο, η πρώτη επίτροπος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και όπως μας είπατε αυτό ε, το χαρτοφυλάκιο ε, θα το μοιραστείτε με τον αρμόδιο επιτρόπο για θέματα ε, μετανάστευσης. Ε, είναι σημαντικό αυτό. Μιλήστε για την ισορροπία, αλλά τα θέματα της ε, διαφάνειας σε περίπτωση κρατήσεις, το PNR, η πρόσβαση στα έγγραψα, ε, τα σκάνερ, ε, τα σωματικά, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και με την ασφάλεια. Στην πρακτική λοιπόν πώς ακριβώς θα συνεργαστείτε με τον συνάδελφό σας, τον Επίτροπο, για να επιλύσετε εφόσον κρυθεί απαραίτητο προστριβές που θα προκύψουν για να διασφαλίζεται το θέμα της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πώς θα μπορέσετε να διαφυλάξετε τα διαφυλάξετε θεμελιώδη δικαιώματα, παρότι δεν υπάρχει σχετική ομάδα εργασία. Και τέλο, όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, πώ ακριβώ ε, προτίθεστε να ενημερώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή την Επιτροπή και πώ τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να διαχυθούν τόσο στην δικαιοσύνη όσο και σε άλλε επιτροπέ. Τρει ερωτήσει κατ' ουσίαν κάνατε και θα πω το εξή. Δέκα χρόνια ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωβουλευτή και είχα επαφές σε μόνιμη βάση με τις επιτροπές. Συνεργαστήκαμε ε, ως ομάδα και αυτό σκοπεύω να συνεχίσω να πράξω και στο μέλλον. Δεύτερον, πώς ακριβώς προτίθεμαι να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου στην ε, Κομισιόν, διότι δεν είναι μόνο η Σεσίλια Μάλστορμ με την οποία θα κληθώ ε, να ανταλλάξω απόψεις. Θα πρέπει να το πράξω και με τους επιτρόπους που θα είναι αρμόδιοι ε, ή την Επίτροπο αρμόδια για τα εξωτερικά θέματα, γιατί όλα αυτά τα θέματα των θεμελιδών δικαιωμάτων έχουν και μία εξωτερική διάσταση. Άρα δηλαδή μιλάμε για διάχυση όλων αυτών των πολιτικών σε πολλού τομεί που είναι πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως υπάρχει ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από τη νέα συνθήκη και το νέο χάρτη και θα βασίζεται επίσης και στο γεγονός ότι η ε, Ευρώπη πρόκειται να ε, συνυπογράψει την ε, συνθήκη θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Θα έχουμε λοιπόν έναν επίτροπο που θα είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όπου υπάρχει κοινή ευθύνη. Παραδείγματο χάρη για τα προβλήματα τα οποία εσείς παρουσιάσατε το PNR, ε, τα SWIFT, ε, τα σκάνερ, τα σωματικά, σωματική πλήρη εξέταση. Ε, μπορείτε λοιπόν να είστε σίγουροι ότι όσον αφορά αυτά τα θέματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία των δεδομένων θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Και επίσης θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις που θα λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε ίσους. Δεν θα δεχθούμε να μας υπαγορεύσουν κανόνες που αντιβαίνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι αντίθετοι οι κανόνες με την προστασία των δεδομένων και αυτά χάρη της επιβολής ε, των κανόνων της τρομοκρατίας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι συζήτησα διεξοδικά με τη Σεσίλια επί του θέματος ε, και υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων ε, και δράσεων. Ο κύριος Μισελ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που σας διακόπτω εδώ, αλλά Ξέρω την εμπειρία που έχετε, τις ικανότητές σας, μας τα έχετε αποδείξει αυτά από τις προηγούμενες θέσεις που κατήχετε. Πάντως για το θεμελιώδη δικαιώματα. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προωθούνται, να γίνονται σεβαστά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε αυτό με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να ελέγχονται και επίσης τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, πώς εφαρμόζουν την ελευθερία του τύπου, τη συγκέντρωση των ε, μέσων ενημέρωσης, την αμεροληψία του κράτους και την βούληση για ε, κυρώσεις έτσι όπως προβλέπονται από τη Νέα Συνθήκη. Ρωτάω λοιπόν, τι συγκεκριμένε πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ή θα μπορούσατε να αναλάβετε προκειμένου τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να τηρούν τις αρχές αυτές, τις οποίες δεν τηρούν όλες οι χώρες μέλη μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνω ότι ο αγώνας που σας περιμένει είναι δύσκολος, σας έχω κάθε εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι εσείς μπορείτε να πιέσετε τα κράτη, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το πώς θα το κάνετε αυτό. Η κυρία Ρέντινγκ να απαντήσει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, βλέπετε, από 1η Δεκεμβρίου, διότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τώρα αποτελεί μέρος της συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αναλύσει κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται προκειμένου να δει κατά πόσο αυθυγραμμίζεται ή όχι με την ε, σύμβαση αυτή. Αυτό όσον αφορά τις αποφάσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή εθνικού δικαίου είναι κάτι που χειρίζεται το δικαστήριο του Στρασβούργου. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνει μέλος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τη στιγμή αυτή και μετά υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Δικαστήριο του Στρασβούργου και το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει να έχει εντολή προκειμένου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ώστε να προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια καλή ισορροπία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα άπαξ και προκύπτει πρόβλημα. Τώρα κατά τα άλλα τι κάνουμε εμείς με τη δικιά μας τη δουλειά. Το ξέρετε κι εσείς από την εποχή που ήσασταν επίτροπος ότι έχουμε αναλύσει όλοι, όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει για να δούμε αν υπάρχει όντως ισορροπία με κύρια οικονομικά ζητήματα. Εφ' εξής, θα αναλύσουμε κάθε πρόταση η οποία βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βλέπουμε κατά πόσο συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι δικιά μου ευθύνη εφόσον αναλάβω τα καθήκοντά μου και συγχρόνως είναι και μια οριζόντια ευθύνη γιατί έχει να κάνει με όλες τις αποφάσεις και με όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφορά επίσης και τις διεθνείς συμφωνίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρωμέβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Ρέντινγκ θέλω εδώ να υπογραμμίσω αυτό που είπατε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια και ελευθερία χωρίς ασφάλεια, αλλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει και ασφάλεια χωρίς δικαιοσύνη. Εδώ δεν μιλήσατε για ελευθερία. Για πείτε μου λοιπόν, τώρα που απειλούνται οι ελευθερίες, πολλές φορές εξαιτία των χειρισμών που γίνονται για να αποφύγουμε τον τρόμο, μπορείτε να μου πείτε εσείς, οι ευρωπαϊκές χώρες περιπτώσεις που είχαμε όπως με τις πτήσεις της CIA ή με τη Swiss την ε, μεταβίβαση δεδομένων, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του ίντερνετ, με τα σκάνερς που βλέπουν ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, εσείς τι θα κάνετε με όλα αυτά. Πώς δηλαδή θα φροντίσετε να είναι ξεκάθαρο, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή των σκάνερς, πώς εσείς θα στηρίξετε τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές όπως είναι αυτή η εξέταση με τα σκάνες. Να απαντήσει η κυρία Ρέντινγκ. Το άρθρο 8 της χάρτας είναι ξεκάθαρο. Τα σκάνες αυτά <clears throat> που βλέπουν την εικόνα στο σώμα του ανθρώπου για να δούνε αν υπάρχει κάποια απειλή, όχι, είναι πράγματα τα οποία βέβαια πρέπει να εξεταστούν με τις εξής ερωτήσεις. Είναι αποτελεσματικά. Ε, δημιουργούν ε, συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο, όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Κάθε φορά που πρόκειται για μια πρωτοβουλία, για μια απόφαση, πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της ε, αναλογικότητας, δηλαδή τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Κάθε μέτρο πρέπει να δούμε αντιστοιχεί στο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. οι ανάγκες μας για ασφάλεια δεν δικαιολογούν κάθε παραβίαση του ιδιωτικού βίου. Οι πολίτες μας δεν είναι αντικείμενα, είναι άνθρωποι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα σκάνερ αυτά. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις σε θελοντική βάση. Πρώτον, δεύτερον, οι εικόνες πρέπει να καταστρέφονται αμέσως μετά. Και τρίτον, πρέπει να ελεγχθούν και οι συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν στην υγεία πρέπει να είναι ασφαλή τα μηχανήματα αυτά. Εξάλλου δεν είναι πανάκια οι, τα σκάνερς αυτά και πρέπει να δούμε και να βρούμε πιο φιλικούς τρόπους να μην παραβιάζει το ιδιωτικό βίος. Και πάνω απ' όλα την αποτελεσματικότητα της συλλογής δεδομένων που έχουμε και το τι χειρισμών τυχαίνουν αυτά. Πρέπει να αξιολογηθούν όλα αυτά για να αποφασίσουμε τελικά για το τι μέτρα ασφάλειας θα παίρνουμε. Είπαμε για το PNR, είπαμε για το SWIFT δεν είναι δυνατόν να καθοδηγούμαστε από τον φόβο, αλλά από τις αξίες πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και γι' αυτό και θα αξιολογείται πάντα με γνώμονα τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε απόφαση και πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τίμωθη Κερκόπ. Ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ παρηγορητικό το ότι έχουμε μπροστά μας ένα άνθρωπο αποδεδειγμένα ικανό. Μιλάμε, Επίτροπε, για μια Ευρώπη 27 χωρών. Με διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας νομοθεσίας και όχι να προσπαθεί να εισχωρεί συστηματικά στις εθνικές δικαιοδοσίες. Η Σύμβαση της Χάγης έχει ακριβώς σαν στόχο όχι τη διεύρυνση του κοινοτικού κεκτημένου, αλλά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Δεν έγιναν πολλά πράγματα. Θα ήθελα να μάθω, Επίτροπε, αν συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέω εγώ, ότι χρειάζονται οι Ευρωπαίοι λιγότερη επιβεβλημένη εκ των άνω εναρμόνιση και περισσότερο συντονισμό. Θα πρέπει να βασιστούμε στα επιτυχημένα στοιχεία του παρελθόντος μας και όχι να εμένουμε σε τομείς τους οποίους δεν θα πρέπει. Κυρία Ρέντινγκ. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το αξιότιμο μέλος. Είμαι πεπισμένη για την εσωτερική αγορά για τα αγαθά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ελεύθερη διακίνηση και τα δικαιώματα των πολιτών. Αν οι κανόνες μας δεν συμφωνούν με αυτές τις δύο βασικές μου πεπιθήσεις, ομολογώ ότι θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες αλλαγές. Αυτό δεν θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο σε εισαγωγικά το λέω αυτό, στον τομέα αν θέλετε του αστικού, στον αστικό ε, τομέα του δικαίου όπου έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Θα είναι όμως πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε άλλους τομείς όπως ε, στο ποινικό δίκαιο. Στον τομέα του ποινικού δικαίου έχουμε συστήματα ενήλικα θα έλεγα με παλιές ρίζες και έχουμε συστήματα επίσης δικηγορικά, δικαστικά κτλ. που εφαρμόζουν τα συστήματα αυτά και που κατανοητά θα προσπαθήσουν να εμείνουν χωρίς αλλαγές στον τομέα τον οποίο γνωρίζουν. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να εμφυσίσουμε εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες του χώρου της δικαιοσύνης έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το νομικό ε, σύστημα να γνωρίζουν ότι και το κοινοτικό νομικό σύστημα είναι κάτι το καλό. Αυτή η αμοιβαία αναγνώριση, αυτή η αποκοινού προσπάθεια θα βοηθήσει. Έχω προσπαθήσει να βελτιώσω το Εράσμους για τους φοιτητές και δημιούργησα επίσης και το Εράσμους Μούντους. Γιατί να μην κάνουμε και ένα Εράσμους για τους δικαστές σαν παράδειγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε επί της ουσίας την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αλλά στον, στον αστικό τομέα δεν υπάρχουν ε, πάρα πολλά προβλήματα και θα προχωρήσουμε θα προχωρήσουμε και με τους ευρωπαϊκούς νόμους όταν οι πολίτες δεν επωφελούνται από την ελεύθερη διακίνηση και με τις διαδικασίες επί παραβάση εφόσον οι ευρωπαϊκοί νόμοι δεν εφαρμόζονται σωστά. Τα βάρες ένα λεπτό. Επίτροπε, αναφερθήκατε στην εποχή που ήσασταν Ευρωβουλευτής. Εκείνη την εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν και τόσο σημαντικό βέβαια όσο είναι σήμερα ενώ είχε λιγότερες αρμοδιότητες. Εγώ είμαι μέλος ε, μόνο εδώ και λίγους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια στιγμή με κάλεσαν για μια συνάντηση που έγινε μια Παρασκευή γύρω από το θέμα της εταιρείας μεταφοράς ε, ε, χρημάτων SWIFT. το SWIFT ε, δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τη βιασύνη την οποία το αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι πάρα πολύ προσεκτικό όταν αντιμετωπίζει τόσο σημαντικά θέματα και να τα συζητά φυσικά αναλυτικά και επιμακρών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στην περίπτωση που έχουμε την δυνατότητα να, να διαπραγματευτούμε εκ νέου εννοώ το θέμα για το SWIFT, τι προτάσεις θα κάνετε. Είδατε κι εσείς ε, πως ήταν τα πράγματα λίγα χρόνια παλαιότερα. Το σύστημα λειτουργούσε εντελώς αδιαφανώς και το Κοινοβούλιο δεν είχε κανένα λόγο. Από την 1η Δεκεμβρίου όμως ε, τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Το Κοινοβούλιο θα έχει λόγο στα πράγματα και ας εξετάσουμε εκ νέου τη συμφωνία για το σύστημα SWIFT έχει συμφωνηθεί για μία περίοδο χρονική μόνο 9 μηνών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την δική του ερμηνεία εννοεί Επίτροπος και τη σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της συμφωνίας αυτής. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να περάσουμε στην διαπραγμάτευση της νέας συμφωνίας για το SWIFT. Και η νέα συμφωνία αυτή για να ισχύσει μετά το πρώτο μήνο θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κανόνες και τις ρήτρε της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε εκεί το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει πλήρως και η Επίτροπος για την Δικαιοσύνη επίσης θα εμπλακεί και αυτή πλήρως. Και όπως σας είπα πριν πάρα πολύ σοβαρά, εγώ θα θέσω τα ερωτήματα όσο δυσάρεστα και αν είναι. Μήπως κάποιες τέτοιες προτάσεις δεν είναι απαραίτητες, μήπως ε, είναι εναντίον ε, του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, μήπως δεν είναι αναλογικές, μήπως είναι κατά των ε, προβλέψεων της, ε, της σύμβασης για τα θεμελιώδη. Εν πάση περιπτώσει εγώ σε συνεργασία με τη Σεσίλια Μάλστρομ και σε συνεργασία με εσάς θα προχωρήσουμε για τη νέα συμφωνία SWIFT. Ε, κυρία Κίνγκα Γκάλ, ένα λεπτό. Μιλάμε για μια νέα εποχή μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και η δημιουργία μιας θέσης όπως αυτήν ε, την οποία καλείστε να καλύψετε είναι μια νέα δυνατότητα, μια νέα ευκαιρία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα στις νέες χώρες μέλη σχετικά ε, με την προστασία των ε, προσωπικών δικαιωμάτων και θα ήθελα εδώ να στρέψετε την προσοχή σας κατά τη διάρκεια της περίοδου που θα είστε υπεύθυνοι στην προστασία των δικαιωμάτων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα εφαρμόσετε τη χάρτα αυτή η οποία είναι νομικά δεσμευτική και πότε θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Για τη χάρτα, καταρχάς λέει η υποψηφία επίτροπος, η χάρτα και ιδιαίτερα το άρθρο 6 όπως είπατε είναι, δεσμευτικά, είναι νομικά δεσμευτικές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της νέας συνθήκης. Νομίζω ότι μπορούμε να νιώσουμε υπερήφανοι για την χάρτα αυτή γιατί δείχνει ότι μπορεί να επιδιώξει κανείς την ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα. Δεν επιβάλλεται εκ των άνω, λαμβάνει σαφέστατα υπόψη τα εθνικά συντάγματα και επίσης την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως επίσης και την πλούσια συλλογή των αποφάσεων της Ολομελίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και όλα αυτά δείχνουν πλέον ότι δια νόμου πλέον αλλά και δια αξιών η Ευρώπη είναι πλέον ενωμένη. Είναι η πιο σύγχρονη κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κόσμο όλο. Δεν το λέμε αυτό δυνατά αλλά έτσι είναι τα πράγματα καλύπτονται και οι πολιτικές ελευθερίες, καλύπτονται οικονομικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα και τα λεγόμενα δικαιώματα τρίτης γενεάς όπως ε, το δικαίωμα ε, σε ε, σωστή και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης, ενημέρωση σωστή από τις κρατικές δομές κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι λόγοι για τους οποίους οι αποφάσεις μας πριν βγουν από την Επιτροπή θα αναλύονται για το κατά πόσον είναι συμβατή με τη συγκεκριμένη χάρτα. Θα υπάρχει μια μελέτη θα έλεγα λοιπόν προκαταρκτική γύρω από τον ρόλο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα εξετάζουμε επίσης και το τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου. Και σε επαναλαμβάνω, θα υπάρξει μηδενική ανοχή σχετικά με την πιθανή παραβίαση της χάρτας αυτής. Σχετικά με τη δική σας εμπλοκή, θα ήταν καλό εφόσον συμφωνείτε να υπάρχει μια αιτήσια έκθεση για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με περιλήψεις των παραπώνων τα οποία εγώ θα λαμβάνω, εσείς θα λαμβάνετε και με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τις οποίες θα θέτετε και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε έτσι και τη σύμβαση αυτή σε σχέση με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις επί τη βάση συγκεκριμένης εντολής το ταχύτερο δυνατόν. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές για τη συμμετοχή της Ένωσης στη Σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ στις ε, απαντήσεις σας αναφέρεστε στην ε, ανάπτυξη μιας χειρής Ευρώπης, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είναι πρώτη προτεραιότητα και λέτε ότι θα ζητήσετε τη βοήθεια ε, του Φορέα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να επιτύχετε την προτεραιότητά σας. Πιστεύετε ότι αυτό προϋποθέτει διεύρυνση αυτού του φορέα. ή μήπως ε, θεωρείτε ότι η διάρκεια ζωής ε, αυτού του φορέα θα πρέπει να πάψει να ισχύει με τη θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Είπατε επίσης ότι ε, βασικό σας καθήκον ε, θα είναι να καταθέσετε και νομοθεσία που να αφορά σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και αυτό τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κράτη-μέλη. Η κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, ο φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, οργανισμός αυτός είναι πολύ σημαντικό εργαλείο διότι αναλύει την κατάσταση που υπάρχει και επιτρέπει σε μας ε, στις αποφάσεις που θα λάβουμε στο μέλλον να έχουμε μια υγιή βάση έτσι ώστε να μην κάνουμε λάθη οποτεδήποτε προτείνουμε αποφάσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για να εξετάσει κανείς το θέμα των διαμαρτυριών, των παραπώνων των ε, πολιτών. Εσείς ως ευρωβουλευτές ε, παίρνετε τις ε, διαμαρτυρίες από την εκλογική περιφέρεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή αν θέλετε η Επιτροπή Αναφορών που είναι μία από τις σημαντικότερες ε, του Κοινοβουλίου. Εγώ υπήρξα πριν από 20 χρόνια πρόεδρος αυτής της ε, Επιτροπής ε, και λοιπόν μπορεί κανείς πραγματικά να κατανοήσει που ακριβώς χτυπάει η καρδιά του πολίτη. Κατόπιν υπάρχει και ο συνήγορος του πολίτη για όλες τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν σχέση με τη διοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα συγκεράσουμε. Υπάρχουν εκατοντάδες διαμαρτυριών που ε, παίρνω και εγώ και οι συνάδελφοί μου οι επίτροποι και αν αναλύσουμε αυτά τα παράπονα μπορούμε να διαπιστώσουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα βασικά προβλήματα και από κοινού πρέπει να έχουμε μια συζήτηση εδώ για να δούμε ε, πού ακριβώς χρειάζεται δράση. Δράση δεν μπορεί να υπάρξει παντού γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει όμως να επιλέξουμε κάποια προβλήματα. Είπα παραδείγματο χάρη ότι επιθυμώ ταχύτατα να προχωρήσω σε θέματα που αφορούν στους εμικτούς γάμους, στην ελεύθερη ε, μετακίνηση κάτω από το πρίσμα της ε, ηθαγένειας, σε θέματα κατω απο το πρισμα της ηθαγενειας σε θεματα διαζυγης ε, παιδιών, ε, βίας κατά των γυναικών. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όπου πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητές μας και μετά από κοινού πρέπει να επιλέξουμε εκείνους τους τομείς όπου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις λόγω αυτών των προτεραιότητων. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σα πω ότι εγώ ανέκαθεν εκτιμούσα ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδεται στο θέμα τη ηθαγένεια. Και όπω ξέρετε, πάνω από το 30% των Ευρωπαίων πολιτών είναι ε, πάνω από 18 ετών και αυτή τη στιγμή η νομοθεσία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα να υιοθετηθεί ε, ένα σχέδιο για τους ανήλικους για να υπάρχει περιθώριο για, τους, ε, για τα παιδιά σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής ε, είναι ένα θέμα, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτυχημένη μάχη κατά αυτών των προβλημάτων. Και η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Ποιε είναι οι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που προτίθεστε να ε, αναλάβετε για να προστατεύσετε τα δικαιώματα των ανηλίκων στη συνθήκη τη Λισαβόνα και στη στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπάρχει επιτέλου μια νομική βάση. Και ερωτώ πώ ακριβώ προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα εκείνα όπου βλέπουμε να υπάρχουν ανήλικοι οι οποίοι είναι αντικείμενο διαμάχης ε, ανάμεσα σε γονείς που χωρίζουν και είναι διαφορετικής ε, ηθαγένειας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει μια νομοθετική πρόταση που θα αφορά τον αγώνα κατά της ε, κακοποίησης, της κακομεταχείρισης και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην πορνογραφία. Η κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, αν δεν ενδιαφερθούμε ή δεν ενδιαφερόμαστε γενικά για τα παιδιά, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Είναι τα πιο ευάλωτα στην κοινωνία μας ε, και χρειάζονται, τη βοήθειά μας πάνω απ' όλα. Ε, για αυτά τα παιδιά κανείς ε, ποτέ δεν μιλάει. Είναι τα αόρατα παιδιά, τα παιδιά που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, τα παιδιά στους δρόμους. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ φέρουμε πραγματική ευθύνη και για το λόγο αυτό θα ήθελα να ενισχύσω τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα παιδιά. Τώρα, συγκεκριμένες δράσεις μου είπατε να αναφέρω και θα τις αναφέρω πολύ σύντομα όσον αφορά την ε, έγκριση, θέσπιση διατάξεων ε, για εγκλήματα κατά των παιδιών. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα συναγερμού διασυνοριακά ή απαγωγή παιδιών από έναν από τους δύο γονείς. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των ε, κρατών μελών. Μία πρόταση που αφορά στο 2011 αφού το 2010 θα έχει προϋπάρξει ανάλυση διότι πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία μέχρι να φτάσουν οι περιπτώσεις αυτές στην τελική τους εκδίκαση στα δικαστήρια και μέχρι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δικαστηριών. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρχει περαιτέρω εναρμόνιση ε, του ε, δικαίου. Κατόπιν Ξέρετε ότι ε, όσον αφορά τις περιπτώσεις διαφορετικών θεγενειών ε, γονέων υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα και θεωρώ ότι δεν μπορούμε πια να περιμένουμε σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση, εμπορία παιδιών. Ε, στο μέλλον θα καταθέσω προτάσεις για την θέσπιση διατάξεων και αυτό σε στενή συνεργασία με την κυρία Μάλστορμ η οποία φέρει και αυτή η ευθύνη για αυτά τα θέματα. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα, εφόσον συμφωνείτε, θα ε, προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τα παιδιά στις διαβουλεύσεις η γλώσσα ε, να είναι φιλική, κατανοητή από τα παιδιά και ελπίζω να με βοηθήσετε εσείς να συμπεριλάβουμε και τα παιδιά σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Ρωμέρο, ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, στη σημερινή κατάσταση με την παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος, εμείς οι πολίτες αντιμετωπίζουμε δύο κάπως αντιφατικές καταστάσεις. Όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα, αλλά συγχρόνως όλοι είμαστε και εν δυνάμει ύποπτοι. Έχουμε ο καθένας το δικό του πορφίλ. Άλλοι είναι μελαχρινοί, είναι από τον Νότο, άλλοι είναι μουσουλμάνοι. Η Ευρώπη δεν έχει αξιοπιστία για να ζητήσει από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, μεγαλύτερο συντονισμό των αστυνομικών και δικαστικών της αρχών. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε εμεί συντονισμό, είναι κάτι που το πληρώνουμε όλοι οι πολίτες. Πιστεύετε λοιπόν ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός πρόληψης του εγκλήματος όπως είναι το Ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Προστασία των Θυμάτων που θα υποβληθεί υπό Ισπανική Προεδρία και μπορεί να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης χωρίς να φροντίσουμε για τον χάρτη πορείας των δικαιωμάτων τόσο των υπόπτων όσο και των θυμάτων με πληροφορίες γιατί εμεί πιστεύουμε ότι πλήττονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι και η βάση της δημοκρατίας. Η κυρία Ρέντιν. Συμφωνώ μαζί σας, απόλυτα. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία στις εξωτερικές μας δράσεις αλλά και στις εσωτερικές μας δράσεις. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος την αρμοδιότητα αυτή την ανέθεσε οριζόντια σε έναν επίτροπο και είπα και στην αρχή ότι θα πρέπει να συνεργαστώ και με άλλους ε, επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για παράδειγμα για τις εξωτερικές σχέσεις. Γιατί οι εξωτερικές μας δράσεις πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο όπως είναι και οι εσωτερικές. Η χάρτα τώρα με όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί πλήρως μέρος της συνθήκης. Αυτό μας ε, δίνει ένα εργαλείο στα χέρια το οποίο δεν είχαμε στη διάθεσή μας νωρίτερα. Τώρα λοιπόν έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και θα τα χρησιμοποιήσουμε, το είπα και στην αρχή, για τις περιπτώσεις εγκληματικών δράσεων, όταν κάποιος είναι ύποπτος, για παράδειγμα. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, θα φροντίσουμε και για τα δικαιώματα των θυμάτων διότι και εδώ χρειαζόμαστε στην πράξη μέτρα. Πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει τα θύματα. Υπάρχουν οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένες χώρες, όχι παντού, και είναι εξοπλισμένοι έτσι που μπορούν να βοηθήσουν. Και ίσως να χρειαστούμε και κάτι πιο ειδικό για την περίπτωση των βιασμών ή της ενδοοικογενειακής βίας. από τη στιγμή που έχει γίνει κάποιο έγκλημα, περνάμε από όλη τη δικαστική διαδικασία και πέρα και από τη δικαστική απόφαση. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά πρέπει να την κάνουμε και σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σόφη Ιντζετφέλτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι μια από τις κύριες ευθύνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι φιλελεύθεροι θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή της. Εσείς όμως ε, βλέπετε κάπως ε, παθητικά και μινιμαλιστικά το θέμα αυτό των ε, δικαιωμάτων, των θεμελιωδών και το αφήνετε περισσότερο στα δικαστήρια και στις χώρες μέλη. Μπορείτε να μας πείτε εσείς πώς θα φροντίσετε για την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τι δράσεις θα πάρετε κατά της ομοφιλοφιλίας, κατά διακρίσεις που γίνονται κατά των θήγων για παράδειγμα ή όσον αφορά τους γάμους μεταξύ ομοφιλόφιλων κλπ. Τι πρωτοβουλίε επίσης θα αναλάβετε προκειμένου να διασφαλίσετε την ελευθερία ε, θρησκείας και ελευθερία συνείδησης. Εσείς θα κάνετε προτάσεις για την εφαρμογή του άρθρου 17 στο διάλογο των εκκλησιών και ε, άλλων οργανώσεων ε, ιδεολογία. Εσείς για θέματα όπως είναι το PNR, το SWIFT και τα λοιπά, τι θα κάνετε εσείς ε, συμφωνήσατε και υποστηρίξατε την μεταφορά δεδομένων προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε τώρα τι θα κάνετε. Η ε, κύριε Ρέντινγκ. Δέκα ερωτήσεις μου κάνατε. Αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Σε μερικές τουλάχιστον. Πρώτον. Όσον αφορά την μεταφορά στοιχείων. Εσείς που είσαστε σε αυτό το χώρο και που συμμετείχετε στην Επιτροπή Ήτρε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσον αφορά την οδηγία για την μη ε, μεταφορά δεδομένων, ξέρετε ποια ήταν η θέση μου. Ήτρα ήταν κατά και το Συμβούλιο Υπουργών Τελεκόμ ήταν κατά. Ε, πρόκειται για ένα Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών που το πέρασε τελικά. Και ελπίζω το Κοινοβούλιο την επόμενη φορά που θα πρόκειται να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα το σκεφτεί δύο φορές πριν πει ναι για μια τέτοια απόφαση. Βέβαια, το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να επαναλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα σε άλλες ερωτήσεις για τη νέα συνθήκη και με ποιο τρόπο από το Δεκέμβριο και μετά πώς ε, θα εξετάζουμε με οριζόντιο τρόπο το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου αυτά να εφαρμόζονται κάθε φορά που έχουμε μια νέα πρόταση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είπα και νωρίτερα, θα εφαρμόζονται και στα κράτη-μέλη κάθε φορά που ένα κράτος μέλος θέτει σε εφαρμογή μία ε, πρόταση ευρωπαϊκού δικαίου. Η ομοφιλοφιλία δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων δεν εξετάζει τον ε, σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει και ο νόμος για το γάμο είναι θέμα των κρατών μελών. Έχει όμως τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει κάθε φορά που ένας πολίτης πάει από μία χώρα σε μια άλλη. Έχει δικαιώματα. Και αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστούμε. Σάμπα Σόγκορ. Θα ήθελα να ρωτήσω τι είδου μέτρα προτίθεστε να λάβετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα τη ε, Στοκχόλμη που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα θα θέσετε τέλο, σε οποιαδήποτε μορφή διακριτική μεταχείριση απέναντι ε, σε ε, αδικήσει βάρο των μειονοτήτων και πώ θα διασφαλίσετε το ότι άτομα που ανήκουν στις παραδοσιακέ εθνικές μειονότητες μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρω προστατευόμενα άτομα όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Η κυρία Ρέντινγκ, και για αυτή την ε, ερώτηση έχουμε δύο νέα στοιχεία στη νέα συνθήκη. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το άρθρο 2 της συνθήκης για πρώτη φορά υπογραμμίζει τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μια μειονότητα. Όχι γενικά σε μια μειονότητα, αλλά τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητα ε, έχουν ε, μεμονωμένα δικαιώματα δικά τους, ατομικά. Υπάρχει λοιπόν στο χάρτη το άρθρο 21 και εγώ προτίθεμαι ε, αυτό το θεμελιώδης δικαίωμα να το υιοθετήσω στην κοινοτική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εκείνης όπου τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. Άρα δηλαδή δύο επίπεδα. Αφενός δημιουργούμε κοινοτική νομοθεσία και δεύτερο επίπεδο τις περιπτώσεις όπου ισχύει η κοινοτική νομοθεσία. Ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα εδώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για να αναλύσει τι ακριβώς διαδραματίζεται και για να μας προσφέρει και τα απαραίτητα στοιχεία. Στη δική μου λοιπόν την ομάδα θα έχω κάποιον που θα είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων. Και ο άνθρωπος αυτός θα είναι απόλυτα αφιερωμένος σε αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή εσείς οι ευρωβουλευτές θα έχετε ε, ένα σημείο αναφοράς. Κάποιον που να μιλήσετε γιατί είμαι σίγουρη ότι εδώ θα έχετε να πείτε πάρα πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να λυθούν αυτά τα θέματα με ένα ιδιαίτερα ρεαλιστικό τρόπο να ε, χρησιμοποιείται η νομοθεσία οποτεδήποτε είναι απαραίτητο και αυτό με βάση τα δικαιώματα που μας αποδίδει η συνθήκη και δίνει τη δυνατότητα ε, να ε, χρησιμοποιηθεί νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το θέμα της ε, ασφάλειας ε, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, είπατε πάρα πολλά και σε σχέση με το SWIFT ε, και βλέπω ότι είσαστε αποφασισμένοι και είπατε και πάρα πολλά για τα σκάνερ ε, σώματος. Ε, κατά την άποψή μου το, ε, το, η συσκευή αυτή πραγματικά είναι κίνδυνος και για την αξιοπρέπεια και για την ασφάλεια του ανθρώπου. Οι δικοί μας λοιπόν οι πολίτες θα περνάνε μέσα από ακτινογραφία και τώρα τίθεται το εξή θέμα. Τα αγαθά όμως, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δεν θα περνάνε μέσα από σκάνερ και ε, από ό,τι γνωρίζετε, ακόμα κι αν ε, περάσει κανείς μέσα από σκάνερ, μετά μπορεί να πάει στο duty free και να αγοράσει πράγματα που δεν το αφαιρούνται. Άρα δηλαδή και εσείς δεν πιστεύετε τελικά αυτά τα σκάνερ σώματος είναι περιτά. Δεν πρόκειται απλά για ε, τυφλές ενέργειας και δεν θεωρείτε ότι πριν εγκατασταθούν τέτοιου είδους μηχανήματα στην Ευρώπη θα πρέπει να εγκριθούν και να εξαστούν πρώτα σε κοινωτικό επίπεδο ή θέλετε το θέμα αυτό να το αφήσετε στα κράτη-μέλη. Η κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, νομίζω τη θέση μου την έχω καταστήσει σαφή όσον αφορά τα σκάνερ σώματος. Όμως αυτά τα σκάνερ είναι ένα μόνο κομμάτι ε, μιας ε, ευρύτερου θέματος. Τα PNR, το SWIFT, ε, όλα αυτά κάποια μέρα θα πρέπει να συζητηθούν και γι' αυτό έχουμε μία σαφή γραμμή επί του θέματος. Ποτέ δεν πρέπει να πανικοβαλόμεθα πρέπει τις αξίες μας επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και που τώρα έχουν καταστεί τμήμα της συνθήκης θα πρέπει αυτές οι αξίες να προβάλλονται ακόμα και όταν διαπραγματευόμεθα διεθνείς συμφωνίες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επαυξάνω. Πράγματι ε, τα ανθρώπινα όντα, οι άνθρωποι δεν είναι δέματα, έχουν αξιοπρέπεια. Και όλα τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν πρέπει πρώτα να διευκρινίζονται. Σέβονται τα μέτρα αυτά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ε, σέβονται το δικαίωμα στην υγεία. Και τα τρία αυτά στοιχεία δυστυχώς ε, δεν εξετάστηκαν. Και τώρα λοιπόν βρίσκονται ε, στην ημερήσια διάταξη. Από κοινού με την κυρία Μάλστορμ θα μεριμνήσω έτσι ώστε τα στοιχεία και τα ερωτήματα αυτά να βρεθούν στο προσκήνιο πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος. Η κυρία Κυρία Επίτροπε, ε, ξέρουμε ότι είστε ε, αποφασισμένοι να προάγετε την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Πώς όμως μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις ε, οδηγίες και τις αρχές περί ισότητας, κυρίως όσον αφορά στους μετανάστες και τους αφήγανους Ρωμά. Παρότι υπάρχουν οδηγίες και κανόνες, ε, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να ασκείται διακριτική μεταχείριση εις βάρος των πλέον ευάλωτων που είναι οι μετανάστες, οι Αθήγανοι Ρωμά, διακοπή από το ακροατήριο. Λοιπόν, ε, το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια οριζόντια οδηγία για την ε, μη διακριτική μεταχείριση. Εσείς τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτό να γίνει νόμος και ε, να ε, μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος όλων αυτών των μειονοτήτων. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν έχω το χρόνο σε δύο μόνο λεπτά να σας ε, εξηγήσω ε, όλα αυτά που έχουν σχέση με την οδηγία ε, περί κατάργησης διακριτικής μεταχείρισης. Και όχι μόνο όσον αναφορά τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους. Έχουμε λοιπόν ε, πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να τα εξετάσουμε. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο διάκειται ιδιαίτερα θετικά απέναντι σε αυτήν την οδηγία και γνωρίζω επίσης ε, ότι εξακολουθούν να εφίστανται ανοιχτά προβλήματα με το Συμβούλιο πρέπει να τα συζητήσουμε διεξοδικά. Από την ερώτηση σας ε, θέλω να διαλέξω κάτι, γιατί είπατε πάρα πολλά, να αναφερθώ μόνο στο, στους Αθήγανους Ρωμά. Κοιτάξτε, υπάρχει μία έρευνα του Οργανισμού περί Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, η μελέτη αυτή υπογραμμίζει ότι οι Ρωμά υφίστανται διακριτική μεταχείριση μια φορά το χρόνο τουλάχιστον όσον αφορά την κατοικία και άλλα παρεμφερή και αυτό δεν είναι αποδεκτό ε, με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ όσον αφορά το θέμα αυτό θα συνεργαστώ στενά ε, με τον Επίτροπο Άντορπ, θα εκμεταλλευτούμε τα διαρθρωτικά κονδύλια που υπάρχουν με καλύτερο τρόπο. Ε, θα εξετάσουμε να δούμε τι ακριβώς λειτουργήσε καλά. Σας ανέφερα το πρόγραμμα Αξεντέρ στην Ισπανία που αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία ε, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να σημειώσουμε και άλλες επιτυχίες. Ε, υπάρχει μια οδηγία περί ισότητας ε, με βάση το φύλλο, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους Αθήγανους Ρωμά. Εγώ θέλω να σας πω ότι η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί για να προκύψουν χειροπιαστά αποτελέσματα ε, θα καταρτιστεί στην Κόρδοβα τον Απρίλιο στη συνάντηση κορυφής με θέμα τους Αθήγανους Ρωμά. Ε, και θα σας συζητήσω και μαζί στα θέματα που πρέπει, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Φαντεκάμπ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ξεκινάει μια περίοδος για συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της δικαιοσύνης και του ποινικού δικαίου ιδιαίτερα. Για αυτά τα θέματα είσαστε πολύ πρόθυμοι για ευρωπαϊκή δράση και εμείς θέλουμε περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες και λιγότερη ελευθερία για τους εγκληματίες. Εσείς μπορείτε να μας δώσετε παράδειγμα τριών συγκεκριμένων πρωτοβουλειών που σκοπεύετε να λάβετε στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης προκειμένου η Ευρώπη να είναι ένας περισσότερο ασφαλής χώρος για τους πολίτες της. Η κυρία Ρέντιν. Νομίζω ότι ήδη το είπα στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Τι δηλαδή πρέπει να γίνει. Πολύ συγκεκριμένα, αλλά και δύσκολα. Γιατί όσο εύκολο μπορεί να είναι στο αστικό δίκαιο να προχωρήσουμε και παρά τα διάφορα στοιχεία τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε αυτό το τομέα, τόσο δύσκολο είναι στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης γιατί εκεί υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Και επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι τα εθνικά κοινοβούλια επίσης έχουν λόγο εδώ. Ένα κράτος μέλος δηλαδή μπορεί να μπλοκάρει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί να προχωράμε προσεκτικά. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Α, έπεσε ο φάκελος για τη δικαιοσύνη. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να πηγαίνουμε προσεκτικά και ότι πρέπει να προσέξουμε πού πάμε. Η αμοιβαία αναγνώριση όμως θα είναι μια τέτοια πρωτοβουλία. Επίσης το εξεκουάτο να καταργηθεί γιατί δεν έχει νόημα. μια ειδική ιδιαίτερη πρωτοβουλία επίσης για το θέμα των τραπεζικών λογαριαζών. Και επίσης το θέμα της ε, Ρώμης 2, το θέμα του να μπορεί κανείς να διαλέξει, είναι κάτι που δεν είναι θετικό και δεν θα είναι δυνατό εφ' εξής. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν πάρα πολύ και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τα κράτη-μέλη και μπορείτε κι εσείς επ' αυτού να βοηθήσετε από τη συνεργασία σας, μέσω της συνεργασίας σας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λαμπρινίδης, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Ρέντινγκ, πριν από ένα μήνα Είπε ένα ε, υπεύθυνο ε, φορέων μετάβαση δεδομένων, είπε ότι δεν έχετε να αποφηθείτε τίποτα από τη μεταβίβαση δεδομένων, άπαξ και δεν έχετε τίποτα να κρύψετε. Ναι, αλλά όποιο δεν έχει τίποτα να κρύψει δεν έχει και ζωή. Όλοι κάτι έχουμε να κρύψουμε εδώ. Ο καθένα μα. Κάτι νόμιμο. Είτε πρόκειται για τι προσωπικέ μα σχέσει, είτε για τι προσωπικέ μα επιλογέ, είτε για τι πεπιθήσει μα, θέματα υγεία. Και από τη στιγμή που όλα αυτά μπουν στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι εμεί συμφωνούμε όλα αυτά να τα κυκλοφορούν και οι διάφοροι φορείς μεταξύ τους. Λοιπόν, εσείς, ως, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008, σκοπεύετε να εξετάσετε και να βάλετε όρια στη συνένεση που θα πρέπει να ε, ζητείτε και να παραχωρείτε από τον κόσμο για να, κυκλοφορεί ευρύτερα, να κυκλοφορούν ευρύτερα δεδομένα για την προσωπική του ζωή αυτή η συναλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, τη συνένεση. Η κυρία Ρέντινγκ. Έχω δουλέψει και συνεργαστεί πολύ με τον Αντιπρόεδρο για τα θέματα αυτά, τότε που συζητήσαμε και αποφασίσαμε για το πακέτο Telecom. Το θέμα αυτό πράγματι ήταν πολύ σημαντικό από τις προτεραιότητές μας δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων θα σας το πω. Μπορεί και να το θυμόσαστε ότι όταν τα δικαιώματα τα οποία ήδη υπάρχουν για τον ιδιωτικό βίο σήμερα δεν γίνονται σεβαστά από μια χώρα, είτε μιας ιδιωτικής οργάνωσης που δρά στο κράτος αυτό, ε, εγώ πήρα τις ευθύνε μου και πήγα στο δικαστήριο στην περίπτωση FORM, P-H-O-R-M, όπου δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς συνένεση. Οι κανόνες είναι σαφείς. Πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει ενημέρωση και συνένεση. Δηλαδή ήδη υπάρχουν σήμερα νόμοι τέτοιοι που εμποδίζουν να γίνεται αυτό που λέτε στο διαδίκτυο. Τώρα η συνάδελφος η Νέλη Κρούς είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα, αλλά επειδή εγώ θα είμαι αρμόδια για τη δικαιοσύνη και εγώ έχω κάποια ευθύνη γι' αυτό, να φροντίζω δηλαδή να υπάρχουν οι σωστοί νόμοι για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους, η οποία προστασία των δεδομένων ρητά αναφέρεται στην νέα συνθήκη. Να ξέρετε ότι εγώ θα φροντίσω για την προστασία των ατόμων. Ευχαριστούμε. Ναταλή Κρίσμπερκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη για τα όσα άκουσα μέχρι τώρα. Σας εύχομαι να τα καταφέρετε στο δύσκολο καθήκον αυτό που θα αναλάβετε και να ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όλο και πιο αποφασισμένο να έχει την Ευρώπη της ελευθερίας και της ασφάλειας. Το είπατε κι εσείς ότι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και, η... και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Αναφερθήκατε και στο άρθρο 6 συγκεκριμένα. Ρωτάω λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς την προσχώρησή μας στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι συμβατό έτσι, ανάμεσα στα όσα περιλαμβάνει η σύμβαση και στις δικές μας τις ρυθμίσεις. Σε θέματα τώρα στικών διαδικασιών, ο πολίτης πρέπει να είναι σίγουρος ότι προστατεύονται τα δικαιώματά του και ότι έχει διαδικασίες και ε, ότι έχει εγγύσει συγγνώμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εσείς τι προτάσεις θα κάνετε και ποια είναι η θέση σας για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Μετά δεν ακούστηκε η ομιλήτρια γιατί χτύπησε το καμπανάκι. Η κυρία Ρέντινγκ. Μπορώ να σας πω πότε θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Πολύ σύντομα, πράγματι. Αμέσως, μόλις, έχουμε την εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, αυτό αναφέρεται στο άρθρο 6 της συνθήκης. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα κατά πόσο το θέλουμε ή δεν θέλουμε, θα το κάνουμε. Και φυσικά και πρέπει να συνεργαστούν τα δύο δικαστήρια. Με ισορροπημένο τρόπο. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαστήριά μας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να τα αποδυναμώσουμε και το δικαστήριο του Λουξεμβούργου πρέπει να παραμείνει αυτό που ήταν όλες αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή να αποτελεί το μέσον, το θεσμό που μας βοήθησε το ευρωπαϊκό δίκαιο να είναι στην υπηρεσία των πολιτών μας και των αγορών μας το ότι συνδυάζονται τώρα τα δύο αυτά δικαστήρια πρέπει να τα ενισχύσει, δεν πρέπει να τα αποδυναμώσει. Δεν θα είναι εύκολο για μας, διότι πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία που πρέπει να επικυρωθεί όχι μόνο από τους 27, αλλά και από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συνεπώς, θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις που μπορεί να αποδειχτούν και δύσκολες, αλλά εγώ, να ξέρετε, ότι θα συνεργαστώ εδώ με τις νομικές μας υπηρεσίες, με το δικαστήριο βέβαια στο Λουξεμβούργο και με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τις Εξωτερικές Σχέσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάσεκ Προτασιέβιτς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κυρία Επίτροπε να θέσω ένα ερώτημα που αφορά στην αποκαλούμενη πρωτοβουλία των πολιτών που εισήχθη με τη συνθήκη της Λισαβόνας και κατά άποψή μου ε, δεν είναι μόνο ένα νέο πολύ σημαντικό θεμελιώδης δικαίωμα αλλά και ένα βήμα ε, να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες καθότι η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο άμεσα στη διαμόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς προβλέπετε ότι θα λειτουργήσει όλο αυτό και πώς ε, ε, θεωρείτε ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί στην πράξη. Η κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο προέκυψε με τη θέση σε ισχύ ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό για να ακουστεί και η φωνή των πολιτών. Μπορεί βέβαια να είναι και επικίνδυνο στοιχείο εφόσον από την αρχή δεν έχουμε ξεκαθαρίσει σε ποια θέματα μπορούν οι πολίτες να λάβουν απάντηση. Παραδείγματο χάρη, αν οι πολίτες μας πούν ότι επιθυμούν να επανέλθει η θανατική ποινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λυπάμαι πάρα πολύ, ε, θεμελιώδη δικαιώματα είναι ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε και με πρωτοβουλία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πριν αυτή η πρωτοβουλία πολιτών ε, εφαρμοστεί στην πράξη πρέπει να διευκρινίσουμε ε, το πλαίσιο, τους κανόνες έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών να εξελιχθεί σε ένα, ένα ιδιαίτερο, ιδιαίτερα θετικό στοιχείο που θα μας δείχνει πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με την τροποποίηση των κανόνων, τη βελτίωσή τους, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία έτσι ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Η δική μου λοιπόν η προσπάθεια θα είναι το συντομότερο δυνατόν να οριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει η πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Και για μένα και για σας όμως είναι πολύ σημαντικό το να μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητες επικοινωνίας έτσι ώστε να εξηγήσω στους πολίτες τι ακριβώς διακυβεύεται. Και για σας όμως είναι σημαντικό ε, το να μπορείτε να ενημερώσετε το, τους εκλογείς σας. Άρα δηλαδή εδώ ε, υπάρχει ε, πεδίο δόξης λαμπρών και για τους δυο μας. Ε, Επίτροπε, έχουμε κάνει ήδη έξι ακροάσεις. Και τώρα θα ασκήσω κάποια κριτική που την είπα και αλλού ότι όσοι και αν ήταν επιτροπή σε όλους ε, μέχρι τώρα τουλάχιστον ε, δεν είχαμε σαφείς απαντήσεις. Εσείς όμως τα καταφέρατε διαφορετικά. Πολύ σίγουροι, πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ε, συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια. Και ε, γι' αυτό ε, προφανώς ήταν και 10 χρόνια επίτροπος, δεν είναι τυχαίο. Τώρα, συγκεκριμένη ερώτηση. Στοκχόλμη και Λισαβόνα και τα δύο αυτά σημαίνουν μεγάλες ευκαιρίες και επίσης ε, σημαίνουν και ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα νέο σύστημα δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν, νιώθετε αισιοδοξία, πιστεύετε ότι τα επόμενα χρόνια θα καταστεί δυνατόν να υπάρχει ένα κοινό δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης κυρία Ρέντινγκ. Έχουμε πολλά δίκαια δικαστικά συστήματα στις χώρες μέλη. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά προσπαθούμε να οικοδομήσουμε στα θεμέλια τα οποία κατά τη διάρκεια των αιώνων έχουν εδρεωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα οι πολίτες μετακινούνται πλέον πάρα σε πολύ μεγάλα ποσοστά από τη μία χώρα στην άλλη. Και υπάρχει μια σύγχυση για το ποια είναι η δικαιοδοσία η κατάλληλη και θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά. Δεν θα πρέπει μόνο να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν τον πολίτη, αλλά θα πρέπει ο πολίτης να είναι πραγματικά ενήμερος για αυτά τα οποία συνιστούν τα δικαιώματά του. Αν αυτός ο οποίος υφίσταται διακρίσεις δεν γνωρίζει τις διακρίσεις αυτές και δεν γνωρίζει συνεπώς τα δικαιώματά του, αυτό είναι μια πολύ αρνητική κατάσταση και πρέπει να ενημερώσουμε σωστά Πρέπει να πληροφορήσουμε και για να το πετύχουμε αυτό μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στον πεδίο του αστικού δικαίου έτσι ώστε να πετύχουμε επίσης την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε αντίστοιχα και σε επίπεδο ποινικού δικαίου, και θα πρέπει οι εθνικοί εταίροι να γνωρίζουν, ε, οι πολίτες της κάθε χώρας να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ε, στην περίπτωση ενός ε, ταξιδιού σε άλλη χώρα, σε περίπτωση εγκατάστασης σε άλλη χώρα, σε περίπτωση ε, ενός διαζυγίου. Όλα αυτά οι πολίτες για όλα αυτά πρέπει να είναι ενήμεροι πρέπει να εφαρμοστούν τα δικαιώματά του. Όποιος δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του δεν τα έχει ουσιαστικά. Για να κλείσει το πρώτο μέρος, Ρωσέτα, ένα λεπτό. Ανάμεσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα πέντε χρόνια είναι και η ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τι θα κάνετε για την δυνατότητα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελία επί τη βάση του Eurojust. Τι θα κάνετε επίσης για τον δημοκρατικό έλεγχο μια ενός τέτοιου οργανισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι προτάσεις θα παρουσιάσετε για, την αμοιβαία, για τον αμοιβαίο σεβασμό των αποφάσεων κατασχέσεων και για την χρήση των κατεσχεμένων αγαθών για κοινωνικούς λόγους και πώς θα διασφαλίσετε την δίκαιη προστασία των συμφερόντων των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε δίκιο ότι η νέα συνθήκη διευκρινίζει ότι βασικός στόχος είναι το Eurojust να μετατραπεί αν θέλετε και να οδηγηθεί σε ένα γραφείο, σε μια υπηρεσία Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Υπάρχουν κάποια εμπόδια, υπάρχουν ε, ερωτηματικά σε επίπεδο οικονομικό σαν παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε ε, αν τα εμπόδια αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, αν τα πρώτα βήματα είναι αρκετά ή αν θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στο μέλλον Όλα αυτά βέβαια άπτονται κυρίως του ποινικού επίπεδου, του πεδίου αν θέλετε και γι' αυτό εδώ χρειαζόμαστε και τη συνεργασία των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Αλλά νομίζω ότι <clears throat> θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια υπηρεσία για την καταπολέμηση του βαρέως εγκλήματος και των, του, σαν παράδειγμα παιδοφιλία, ένα φαινόμενο, ένα παράδειγμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα. Εκεί θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία την οποία έχουμε για να βρούμε τις λύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την καταπολέμησή τους. Στο ποινικό πεδίο υπάρχουν πάντα δύο στοιχεία. Υπάρχει το στοιχείο αυτού ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα ή υποτίθεται εν πάση περιπτώσει ότι το έχει διαπράξει και αυτός έχει κάποια δικαιώματα βέβαια και στην δημοκρατία θα πρέπει εμείς να δώσουμε εγγυήσει για τα δικαιώματα αυτά μέχρι ότου καταδικαστεί. Και αυτή τη στιγμή καταδικαστεί και φυλακιστεί και εκεί έχει κάποια δικαιώματα και αυτά θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από την άλλη έχουμε εκτός από τους θύτες τα θύματα. Δεν θα πρέπει εμείς ε, να κοροϊδεύουμε ε, τα θύματα ότι τα βοηθάμε. Παράλληλα με τα συστήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών οι οποίοι έπεσαν θύματα κάποιων εγκληματικών ενεργειών, κάτι το οποίο ποτέ δεν επεδίωξαν. Όχι, όχι διακοπές. Μια κυρία από το κοινό η οποία όμως δεν ακούγεται. Please. Ε, δεν σας δίνω το λόγο λέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ είστε ευγενείς και σεβαστείτε τους κανόνες όπως όλοι. Ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ και τα μέλη για τη συνεργασία και την κατανόηση την οποία έδειξαν. Θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα των ερωτήσεων να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής των Δημοσίων Ελευθεριών ότι θα γίνει μια αξιολόγηση των απαντήσεων στις 6 και θα προηγηθεί συνάντηση των συντονιστών της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών στις 5 και μισή.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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass... Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, ε, παρακαλώ ε, αργά αλλά σταθερά να ξαναπεράσουμε σε επίπεδο ακρόασης. Ich denke, wir werden das auch recht zügig machen, einen geschäftsleitenden Hinweis zu Beginn. Εκείνο μπορούμε να τελειώσουμε και γρήγορα. Ε, να σας πω το εξής, μας ενημέρωσαν ότι έχουμε 30 Α, μπορούμε να δουλέψουμε, να παραμείνουμε άλλα 30 λεπτά, να διαρκέσει η ακρόαση 4 ώρες. Που σημαίνει ότι οι συνάδελφοι ε, μπορούν να μιλήσουν όσο θέλουν και όσοι θέλουν και δεν θα υπάρχει περιορισμός. Κατά τα άλλα, θα είμαι σύντομος ε, στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Ε, να σας πω ότι η διαδικασία θα είναι λιγάκι διαφορετική σε αυτή την Επιτροπή. Με την έννοια ότι όσοι κάνουν ερωτήσεις έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν για ένα λεπτό μετά η Επίτροπος ε, θα απαντήσει για δύο λεπτά και κατόπιν υπάρχει και η δυνατότητα συμπληρωματικής ερώτησης. Αλλά παρακαλώ για το ίδιο θέμα, όχι για άλλο διαφορετικό θέμα. Και κατόπιν ε, η Επίτροπος ε, θα κληθεί τη συμπληρωματική ερώτηση να την απαντήσει μέσα σε ένα λεπτό. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην Νομική Επιτροπή. Κυρία Επίτροπε που είσαστε υποψήφια για θέματα δικαιοσύνη. Σας καλωσορίζω και ευθύ εξ αρχή. θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να κάνετε τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, στη δική σας Επιτροπή θα συζητηθούν τα θεμελιώδη νομικά προβλήματα της Ένεσης. Αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και σε επίπεδο αστικό και σε επίπεδο εμπορικό και σε επίπεδο νομολογίας. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι δικηγόρος και θαυμάζω τις νομικές σας γνώσεις και γενικότερα την εμπειρογνωμοσύνη σας στον συγκεκριμένο τομέα και γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας χρησιμοποιήσω όσο περισσότερο μπορώ τα επόμενα χρόνια. Είμαι πολιτικά δραστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια, πρώτα σαν Ευρωβουλευτής και μετά σαν Επίτροπος. Έχω λοιπόν μια κάποια εμπειρία και γνωρίζω τη σημασία που έχει ο νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο υπερεθνικός, ε, η υπερεθνική νομική τάξη θα έλεγα βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση αυτή δεν ε, αποτελείται από δυνάμεις ασφαλείας μόνο ή από το δικαστικό σώμα ή τους στρατιωτικούς, αλλά από την πεποίθηση την οποία όλοι έχουμε ότι ο νόμος θα πρέπει να γίνεται σεβαστός, να εφαρμόζεται και ε, όπως είπε ο Βάλτερ Χάλσταϊν, απαιτείται μια κοινότητα η οποία να βασίζεται στην, στο κράτος του δικαίου, στην τάξη του δικαίου. Αυτή η κοινότητα του δικαίου, αυτήν χρειαζόμαστε. Έχουμε πολλά πετύχει μέχρι τώρα. Έχουμε μια ιστορία στον τομέα αυτό παρά τις διαφορές μας και οι Ευρωπαίοι κατάφεραν μέσα από τις διαφορές αυτές να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις και σε συγκεκριμένα βήματα προόδου. Ενότητα αλλά από την άλλη και ποικιλία Έχουμε εντελώς διαφορετικές παραδόσεις κάποιοι από εμά, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ένα υπερεθνικό σώμα δικαίου το οποίο είναι χρήσιμο για όλους. Έχουμε μάθει ε, σύμφωνα με αυτό να ακούμε ο ένας τον άλλον, να συγκρίνουμε τα συστήματά μας και να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε ένα ισχυρό κοινοτικό νομικό σύστημα. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει ο νόμος να είναι πάντα η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα προτείνει, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα σχολιάζει και θα τροπολογεί και εμείς θα είμαστε στη θέση που βρισκόμαστε για να ελέγξουμε και το σεβασμό του δικαίου και φυσικά αυτό θα γίνεται εν πλήρη σεβασμό των εθνικών νομικών παραδόσεων. Το έχω πει αυτό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στον ποινικό τομέα όπου η συνεργασία μας είναι θα έλεγα σχετικά πρόσφατη όπου τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν ένα σημαντικό λόγο και στον τομέα του ποινικού είναι σαφές ότι θα πρέπει να προκαλέσουμε μια κάποια νέα συνένεση. Στο αστικό πεδίο και στο εμπορικό πεδίο θα συνεχιστεί η συνεργασία, θα εμβαθυνθεί και όπου απαιτείται να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Πάντα στον τομέα τον αστικό και τον εμπορικό θα πρέπει να είμαστε και μπορούμε νομίζω να είμαστε φιλόδοξοι γιατί ακριβώς με βάση τις ρυθμίσεις αυτές τις νομικές οι επιχειρήσεις μας μπορεί να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν σε επίπεδο γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα επιχειρήσεις οι οποίες ε, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλές χώρες. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει επίσης και για την έξοδο από την οικονομική κρίση, γιατί η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς είναι ο καλύτερος τρόπος για μια σωστή ανάκαμψη οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η εσωτερική αγορά σαφώς και μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Γνωρίζω τις πρωτοβουλίες, τις εκθέσεις πρωτοβουλίας τις οποίες έχετε υπερψηφίσει και ζητείτε να υπάρξουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κάποιες από τις προτάσεις αυτές ε, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές και θα προσπαθήσω να τις προωθήσω εφόσον με επιλέξετε. Γιατί έχει απόλυτα ε, νόημα οι προτάσεις σας. Η κατάργηση του εξεκουάτου σαν παράδειγμα η οποία κοστίζει από 800 με 2.000 ευρώ σε αμοιβέ δικηγόρων και νομικών συμβούλων σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται βέβαια κάποιες ε, ρυθμίσεις, κάποιες προφυλάξεις. Η κατάργηση όμως του εξεκβάτορη είναι σίγουρα μία πρώτη λύση. Δεύτερον, υπάρχει μία πρόταση Έξι λεπτά κανονικά έπρεπε να είχατε μιλήσει. Θα είμαι πολύ συνοπτική από εδώ και πέρα, λέει η κυρία Ρέντινγκ. Οι ευθύνε στα ατυχήματα τα οδικά, σαν παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτές. Υπάρχουν 500.000 ατυχήματα κυκλοφορίας σε αιτήσια βάση. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ομοιογενούς αντιμετώπισης Πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση Απαιτείται να υπάρξει επίσης συμβατότητα ανάμεσα στις συμβατικές ρυθμίσεις σε επίπεδο συμβάσεων και όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, λέει συνοπτικά η Επίτροπος, με σωστή και ισορροπημένη αντίληψη, προστατεύοντας και τα δικαιώματα των καταναλωτών Το κοινό πλαίσιο αναφοράς επίσης, το λεγόμενο πολιτικό κοινό πλαίσιο αναφοράς στο CFR, σίγουρα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό, πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Είναι θα έλεγα το έμβριο και για έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα. Εν πάση περιπτώσει θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Θυμίζω εδώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκίνησαν με ένα ενιαίο εμπορικό κώδικα. Γιατί να μην υπάρχει ένας αντίστοιχος αστικός για τη λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι σας ακούω πάρα πολύ ευχάριστα, ε, δεν τη θέμα από αυτού και λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να σας διακόψω. Συνεχίζουμε όμως τις ερωτήσεις και το λόγο έχει ο κύριος Αντέος από το ΕΛΚ για να υποβάλει την ερώτησή του. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για αυτή την δήλωση. Ευχαριστώ για αυτό το οποίο είπατε, ότι κάποιες από τις προτάσεις μας και τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες ε, θα προσπαθήσετε να τις κάνετε πραγματικότητα και θα σας βοηθήσουμε. Ξέρετε ότι στο τέλος του 2009 το Κοινοβούλιο είχε κάνει κάποιες προτάσεις για, τα, για τις νομικές ρυθμίσεις γύρω από τον γάμο και για κάποιες διαδικασίες που αφορούν επίσης ε, και τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία μέσα από το γάμο όπως επίσης και τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, είχατε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποιες προτάσεις στην αρχή της ε, περίοδου της ανάληψης εντολής την οποία θα έχω. Είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση την οποία αυτή για μας και καλό θα είναι το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσετε γιατί έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο στο Συμβούλιο γύρω από τα θέματα του γάμου. I do not like when Europe advances. Η Ευρώπη πράγματι όταν προχωρά μέσω των μορφών ενισχυμένης συνεργασίας δεν μου αρέσει. Όταν κάποιες χώρες προχωρούν και όχι όλες μαζί ε, με στεναχωρεί. Κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό θα φροντίσω έτσι ώστε και οι 27 χώρες να προχωρήσουν μαζί. Όταν βλέπω όμως ότι σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως η Ρώμη 3 δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με ομοφωνία τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην υπάρχουν άλλες δυνατότητες παρά να προχωρήσουμε. Ξέρετε τα στοιχεία και τους αριθμούς. Έχουμε 350 μικτούς γάμους. Κατέτος στην Ευρώπη 350.000 και 170.000 μεικτά διαζύγια. Δηλαδή το 20% του συνόλου των διαζυγίων αντιπροσωπεύουν ε, διαζύγια μεικτών γάμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προβλήματα δημιουργούνται επίπεδα γαμικών συμβάσεων, προβλήματα για τα παιδιά αυτών των ενώσεων. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες έστω και μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Δέκα χώρες το έχουν ζητήσει αυτό και θα πρέπει να προχωρήσω. Ελπίζω εν τω μεταξύ όταν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δουν ότι είμαστε πραγματικά αποφασισμένοι να μας ακολουθήσουν, να μας συνοδεύσουν και αυτό έχει μεγάλη σημασία για να μην είμαστε μόνο 10 αλλά έστω και 20 και 27 στο τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Herzlichen Dank, Herr Kollege Nachfrage bitte ερώτηση παρακαλώ. Κοιτάξτε, δέκα χώρες ζήτησαν αυτή τη ε, διαδικασία την ε, ενισχυμένη και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσείς ε, προβλέπετε να εισάγετε τροποποιήσεις στην αρχική σας πρόταση. Κοιτάξτε. Αυτή είναι μία από τις προσπάθειες τις οποίες θα κάνω εφόσον αποφασίσετε ότι θα είμαι επίτροπος. Μέχρι τώρα έχω ασχοληθεί όπως πρέπει άλλωστε με τα γενικά και δεν μπορώ να περάσω σε λεπτομέρειες αλλά έχει ήδη υπάρξει προπαρασκευή δεν έχουμε μπροστά μας κάτι το καινούριο και επί τη βάση αυτής της παρασκευαστικής εργασίας θα ζητήσω από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εμπειρία γύρω από τα θέματα αυτά να μου δώσουν τις απόψεις τους, να μου μεταφέρουν τις απόψεις τους έστω και ανεπίσημα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα με βοηθήσει, θα με βοηθήσει <laughs> συγγνώμη. Αλλά θα ήθελα για τέτοιες σημαντικές αποφάσεις ε, να μην καθυστερήσουμε. δεν θα πρέπει να ε, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, η ασθενής πλευρά ε, σε τέτοιου είδους καταστάσεις και σίγουρα αυτό απάρει της εικόνας που έχω εγώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ραπκάη. Κυρία Ρέιντινγκ, στην γερμανική εφημερίδα Die Welt χτες σας περιέγραψαν ως την ε, γυναίκα που έχει γοητεία, που έχει γνώσεις, αλλά και τη γυναίκα εκείνη η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ε, στις επιχειρήσεις. Γιατί, γιατί ε, υπάρχει η άποψη ότι θα έχετε να κάνετε και με επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν αναφέρεται στην ε, εφημερίδα ότι δεν θα πολεμήσετε και δεν θα παλέψετε για την αντιμετώπιση και κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης. Αυτά είναι αρμοδιότητες άλλων επιτροπών, αλλά και εμείς είμαστε αρμόδιοι για την προστασία του καταναλωτή, ε, για τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων και έχοντας κατά νου την ευρωπαϊκή ιδιωτική επιχείρηση, εκεί υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα που αφορούν στη συναπόφαση. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να μου πείτε, αυτά που διάβασα με φόβησαν λιγάκι. Μπορείτε εσείς να με καθησυχάσετε και ανέμε ναι, με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, ως πρώην δημοσιογράφος ε, ποτέ δεν θα τολμούσα ε, να σχολιάσω τη δουλειά ενός πρώην συναδέλφου. Αν όμως αυτός ο ή η συνάδελφος είχαν απευθυνθεί σε εταιρείε στον τομέα των τηλεοπικοινωνιών δεν θα έπαιρναν ε, την ίδια απάντηση. Α πάρουμε παραδείγματο χάρη το θέμα τη περιαγωγή. Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε εκεί. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανεί υπέρ ή κατά και αυτό κατηγορηματικά. Ε, να αναζητά κανεί ισορροπίε. Έχουμε την ισόρροπη αγορά με το δικαίωμα τη ελεύθερη μετακίνηση για του πολίτε. Έχουμε επίση και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα μη διακριτική μεταχείρισης έναντι των πολιτών. Μπορούμε λοιπόν να επιτύχουμε την ισορροπία. Και εγώ είδα σε κάποια γερμανική εφημερίδα που την έχω και κάπου μαζί μου μάλιστα, εκεί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ανάλυση ενός γερμανικού πανεπιστημίου που καταλήγει στο ότι σε εκείνες τις επιχειρήσεις όπου υπάρχει αρκετά υψηλή απορρόφηση γυναικών, αναπήρων και όπου υπάρχει και διακριτική μεταχείριση εις βάρος ανθρώπων, αυτές οι επιχειρήσεις τελικά τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ισορροπία στην κοινωνία μας που πρέπει να διατηρηθεί μερικές φορές. Πρέπει κανείς να ε, πλησιάσει περισσότερο τις επιχειρήσεις και άλλες πάλι περισσότερο τους καταναλωτές. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι στην ε, ε, οδηγία για τον καταναλωτή θα λάβω πλήρω υπόψη μου τα θέματα της προστασίας ε, του καταναλωτή. Ξέρω πολύ καλά την κριτική που έχει ασκηθεί και μπορώ να σας πω το εξής. Αν τελικά την οδηγία για τον καταναλωτή, εάν εκεί διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν απάτες, ξεχάστε την. Άρα δηλαδή πάντα πρέπει να αναζητούμε ισορροπίες ανάμεσα σε διαφορετικά συμφέροντα και εγώ, πιστέψτε με, θα το παλέψω. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε αυτό με την γοητεία και την επιμονή. Ισχύει, το διαπιστώνω και εγώ, η διεισόμαση, αλλά επανέρχομαι στα θέματα κατανοητή που τα θίξετε κι εσείς. Δηλαδή, ε, δεν είναι ότι πρέπει μόνο να προστατεύουμε τα δικά τους ε, τα δικαιώματα, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον ε, θέλουμε να επιτύχουμε εναρμόνιση προς τα κάτω ή προς τα πάνω, προς το ελάχιστο ή προς το μέγιστο. Και εδώ και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει διάσταση απόψεων και θα ήθελα να μάθω τη δική σας την άποψη. Ε, θέλω να σας πω ότι ως Επίτροπος για θέματα τηλεπικοινωνιών τα τελευταία πέντε χρόνια και επίσης και ως Επίτροπος αρμόδια για θέματα διασυνοριακών αγορών μέσω του ίντερνετ. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ότι με την, με την εναρμόνιση προς τα κάτω ποτέ θα μπορέσουμε να πετύχουμε την κοινή αγορά. Το θέμα δεν είναι οι διασυνοριακές επιχειρήσεις να νορμονιστούν προς τα κάτω. Γιατί έτσι ποτέ κανείς δεν θα επιτύχει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ποτέ αυτοί δεν θα θελήσουν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους. Βλέπουμε ε, για την οδηγία ε, οι αγορές για το online δεν αναπτύσσονται πλήρως γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι <clears throat> η εναρμόνιση προς τα πάνω είναι η απάντηση και γνωρίζω επίσης ότι πρέπει να δούμε λιγάκι την ποιότητα ε, του σχεδιασμού και της ε, προστασίας. Θα το εξω αυτό όταν ε, θα το ερευνήσουμε με τους νομοθέτες και θα βρω από κοινού με εσάς και με το Συμβούλιο πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Μπαλτασάρα. Μας είπατε κυρία Ρέντινγκ ότι μία από τις προτεραιότητές σας είναι η δημιουργία της Ευρώπης των πολιτών. Συνεπώς έχετε την πρόθεση να ξεκινήσετε λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα που θα οδηγήσουν στο να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Μετακινήσεις, ε, διαπροσωπικές σχέσεις, εμπορικές συναλλαγές. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Για να είμαστε σίγουροι για τον σεβασμό των διαφορετικών νομικών πολιτισμών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αμοιβαίας αναγνώρισης οι αυθεντικές αυτές ε, ε, πράξεις δεν λαμβάνονται και δεν εκδίδονται μάλλον σε όλες τις χώρες στο ίδιο επίπεδο, σαν παράδειγμα από συμβολιογράφους. Μήπως ε, λοιπόν αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να μην καλύψουμε σε μια πρώτη φάση στα πλαίσια της αμοιβαία αναγνώρισης στα συμβολιογραφικά, αλλά να επεκταθούμε και σε άλλες νόμιμες, σε ορισμένες χώρες πράξεις. Ναι. Αυτά είναι πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, βέβαια, αν διαβάσετε την έκθεση Λαμασούρ θα δείτε πάρα πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα του γιατί δεν δουλεύει. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε λύση για αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια πιο οριζόντια αντιμετώπιση της αμοιβαία αναγνώρισης. Σήμερα έχουμε μια αναγνώριση και ξεκινάμε και με τον συνάδελφο που είναι τώρα επίτροπος ξεκίνησε με τα κληρονομικά δικαιώματα τα διασυνοριακά είναι νομίζω ένας καλός τρόπος να προχωρήσουμε και εγώ βέβαια θέλω να προχωρήσω ακόμα περισσότερο και για όλα τα άλλα. Όχι όμως από πάνω προς τα κάτω. Θέλω πρώτα μια δημόσια διαβούλευση για όλα αυτά τα ζητήματα προκειμένου να μάθω από τους πολιτικούς, από αυτούς που αποφασίζουν, αλλά και από τους πολίτες και από τους διάφορους κλάδους να μάθω τι χρειάζεται και από τους επαγγελματίες φυσικά που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση και μετά να οδηγηθώ σε μια συγκεκριμένη δράση. Συμπληρωματική ερώτηση. La soluzione potrebbe essere... Κοιτάξτε, η λύση θα μπορούσε να είναι να υπάρχει ένας οργανισμός ευρωπαϊκός ο οποίος θα εγγυάται την νομιμότητα αυτών των πράξεων. Ε, δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί ένας ε, κοινό ε, παρανομαστής για την αυθεντικότητα όλων αυτών των εγγράφων. θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Είναι μία αυτή μεταξύ πολλών δυνατοτήτων. Ίσως να μην πρέπει να υπάρξει ένας νέος θεσμός. Εγώ βλέπετε δεν είμαι και πολύ υπέρ του να δημιουργούμε νέες δομές. Σίγουρα όμως θα το κοιτάξω αν μπορεί να γίνει με κάποιο θεσμό που ήδη υπάρχει και εύκολα στην πράξη, τόσο το καλύτερο. Πάντως ακριβώς γι' αυτό και την χρειαζόμαστε την δημόσια διαβούλευση, ώστε να ακουστούν οι διάφορες ιδέες, να τις αναλύσουμε να δούμε πόσο εφικτές είναι και τι δυνατότητες υπάρχουν εφαρμογή τους στην πράξη. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους εκείνους που εξέφρασαν σεβασμό για το έργο σας στην Κομισιόν ιδιαίτερα όταν ασχοληθήκατε με το πακέτο τηλεπικοινωνιών, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Η ανακοίνωση του Οκτωβρίου του 2009 λέει ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια φιλόδοξη ε, πρωτοβουλία για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εσείς λοιπόν πώς βλέπετε το ρόλο σας ως επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια στα πλαίσια των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και πώς θα φροντίσετε να υπάρξει ισορροπία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την ελευθερία. Ένα γαλλικό δικαστήριο έχει πει ότι πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο τελικά υπάρχει περιθώριο για νέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πάνω απ' όλα για να δούμε πώς θα τα θέσουμε σε εφαρμογή. Και συγκεκριμένα για τα δικαιώματα, τα πνευματικά των συγγραφέων στα πλαίσια του διαδικτύου. Και τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για την εφαρμογή όλων αυτών. Η κυρία Ρέντινγκ, όλη αυτή η συζήτηση για το copyright έγινε και ξανάγινε στο σώμα. Και ξέρετε ότι εγώ υποστήριξα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άρθρο 138 όσον αφορά τις νέες ελευθερίες στο ίντερνετ. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση, αλλά τα καταφέραμε να περάσει τελικά ε, με συνδιαλλαγή στο Συμβούλιο. Αυτό συμβαίνει ότι αυτές οι νέες ε, διατάξεις ελευθερίας στο διαδίκτυο ενισχύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτή βέβαια είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι δημιουργοί πληρώνονται για το έργο του. Από τη συζήτηση φάνηκε ότι δεν μπορεί να βρούμε λύση με τα μέσα που είχαμε στον παλιό κόσμο. Ότι χρειαζόμαστε νέα, πιο σύγχρονα μέσα για να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία και τη δημιουργία. Πάντα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ε, προστασία, νομική προστασία και διασυνοριακά. Με την προσφορά και όχι με την καταστολή, γιατί καταστολή δεν έχει νόημα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ήταν ξεκάθαρο με την απόφαση αυτής, συναπόφαση απόφαση δηλαδή για το πακέτο Telecom, ότι νόμοι όπως αυτός που προτάθηκε στη Γαλλία δεν θα αποτελέσει ποτέ μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου. Συμπληρωματική ερώτηση θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία, μια διεθνή συμφωνία κατά της παραποίησης. Εσείς τι γνώμη έχετε για τη συμφωνία αυτή. Εσείς πιστεύετε ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει διατάξεις με κυρώσεις Ακόμα και αν πρόκειται για εμπορικού σκοπού. Εσεί στην περίπτωση τη Γαλλία είπατε ότι αυτή η γαλλική επιλογή δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή επιλογή και ότι πρέπει να βασιστούμε σε κάτι άλλο. Η κυρία Ρέντινγκ, όπω ήδη εξήγησα στη συζήτηση εδώ πολλέ φορέ, το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνθήκη της έχει ανθρώπινα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χάρτα θεμελιδών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι κάθε απόφαση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περνάει πρώτα από μία αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι οριζόντια ευθύνη αυτή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι και όταν πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες, για τις επόμενες δηλαδή, που θα εξεταστούν και από το δικό σας σώμα εννοείται, αυτό το θέμα θα ληφθεί υπόψη με ψηλή προτεραιότητα. Για τα θέματα ποινικού δικαίου, για τα πλαστά προϊόντα, με την συνάδελφό μου, τη Σεσίλια Μάστρομ, θα εξετάσουμε κυρώσεις για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται για το downloading, έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό, τα πλαστά προϊόντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο άλλο τα παραπημένα προϊόντα και άλλο το downloading που γίνεται στο διαδίκτυο. Πολλές φορές θα μας δοθεί ευκαιρία να ψάξουμε να βρούμε ισορροπία ανάμεσα σε δύο δικαιώματα. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας από τη μία και το δικαίωμα της ε, ιδιοκτησίας της ε, του έργου, της δημιουργίας. Η δημιουργία από τη μια και η διοκτησία από την άλλη. Πράγματι είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς τόσο επίμαχα θέματα σε σύνομο χρονικό διάστημα, ε, όμως και εμείς κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η κυρία Γόλης. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία ε, επίτροπε υποψήφια ε, για τις αρμοδιότητες που γνωρίζουμε. Μας δώσατε πράγματι ένα, μια πολύ ένα πολύ εντυπωσιακό δείγμα αυτό που θα ε, πράξετε στο θέμα των ε, ελευθεριών του πολίτη. Το θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Εγώ ανησυχώ για το κατά πόσο θα μπορέσουμε τελικά να κατανοήσουμε και να ε, περάσουμε προς τα έξω ένα προσπελάσιμο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε 27 ε, διαφορετικές νομοθεσίες, ε, διαφορετικές ρυθμίσεις και πολύ σωστά λέτε ότι εσείς θέλετε να προχωρήσετε παραδείγματος χάρη στα, στα πρωτότυπα έγγραφα, στις διαθήκες ε, στην Αγγλία, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν ε, δυσκολίες λόγω του εθνικού δικαίου. Ως εκ τούτου υπάρχουν ε, πολλοί πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τι θα κάνουμε τελικά. Θα είναι το σύστημα προσπελάσιμο για τους πολίτες και θα μπορεί να ταυτιστεί με, την, με τα δικαιώματα των πολιτών. Κοιτάξτε, η κυρία Αντιπρόεδρος, ε, εσείς κυρία Γόλη, ε, θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων θα έλεγα. Και είπα και προηγουμένως ότι η δικαιοσύνη υπάρχει μόνο εφόσον γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και ένας από τους τρεις ε, πολίτες σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος δεν γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κενό και εδώ πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Γνωρίζω λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει πρόοδο στο θέμα αυτό. Ε, το εξέτασα από κοινού ε, με την υπηρεσία ε, δημοσιοποιήσεων, δημοσιεύσεων ε, που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και θέλω να σας πω ότι η εθνική δικαιοσύνη, οι εθνικές νομοθεσίες ε, θα είναι διαθέσιμες, θα υπάρχει μία περίληψη έτσι ώστε τα πράγματα να είναι πιο απλά. Πάντως, σας λέω, αυτά είναι στη φάση της διεργασίας. Θα υπάρχει ε, μία ε, ενιαία πύλη το 2011. Επίσης, ε, γνωρίζετε ότι δουλεύουμε και για την ε, ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Για αυτή την πύλη ξεκινήσαμε το 2006, το 2007, δεν θυμάμαι ακριβώ, ε, θα έλεγα το 2007 μάλλον, και τότε είχαμε την πρώτη επεξεργασία το 11 και το 14 θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πύλη από όπου ε, θα μπορεί κανείς ε, να αποκομίσει αντιδράσεις, ε, να αποκτήσει τα έγγραφα, να έχει την πιστοποιημένη υπογραφή. Θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά. αυτά αυτές είναι οι πύλες. Τα άμεσα αποτελέσματα για το όταν επιθυμεί κανεί ένα έγγραφο το πώς ακριβώς μπορεί να το αποκτήσει πολύ συγκεκριμένα αυτά θα τα συζητήσουμε κάτι άλλο σημαντικό είναι να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες για τα δικαιώματά τους εδώ τίθεται πραγματικά το θέμα της ηθαγένεια, που ε, με αφορά εμπίπτει στι δικέ μου αρμοδιότητες νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν ως εργαλείο για να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. Και εδώ λοιπόν χρειάζομαι τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί και εσείς ε, πρέπει να ενημερώσετε τους ε, πολίτες για τα δικαιώματά τους. Και υπάρχουν πολλοί πολίτες ε, που ταξιδεύουν, ζουν στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν εκεί προβλήματα και επιθυμούν μια λύση. Θέλουμε και αυτούς να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ε, δεν έχω πρόβλημα αυτά που είπατε για την επικοινωνία και συμφωνώ, αλλά ε, δεν απαντήσατε σε κάτι άλλο που έχει σχέση με την ερώτησή μου. Δηλαδή, ακριβώ λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετικέ μέθοδοι προσέγγιση και υπάρχουν και διαφορετικέ απόψει για την ενισχυμένη συνεργασία, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ε, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα μείνει εκτός της ε, προστασίας ε, με πολιτικά ε, δικαιώματα, με δικαιώματα του πολίτη. Τα Ιωνί είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από ποτεδήποτε στα 11 αυτά χρόνια που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είπατε μόνοι σας. Η δυνατότητα να υπάρξει ένα σύστημα των 28 ή ένα σύστημα το 28 που θα επιβληθεί στα 27, αυτό ε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Είναι βέβαια και μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Όμως αυτή η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, τρέχει αυτή η συζήτηση, διεξάγεται και όπως είπα στην ε, εισαγωγή μου, εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Εγώ θέλω να ακούσω την άποψη όλων των δικηγόρων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και που συνεργάζονται μαζί σας, γιατί θα με βοηθήσει αυτό έτσι ώστε να καταλήξει η Επιτροπή σε μια ικανοποιητική λύση. Μπορώ να σας πω ότι στη Γενική Διεύθυνση, όπου ελπίζω να δουλέψω, εφόσον με εγκρίνεται, υπάρχει πληθώρα ε, καλών δικηγόρων πάρα πολύ καλή δικηγόροι και στο δικό μου το ιδιωτικό γραφείο. Νομίζω λοιπόν ότι θα βρούμε τελικά τη λύση εκείνη που θα είναι και η καλύτερη για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων ε, που ε, ζουν σε χώρα όπου ισχύει η νομολογία. Η νομολογία εξάλλου είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σεβαστό και δεν πρέπει να την αγνοούμε. Ο συνάδελφος κ. Μποντό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας για τον Ευρωπαϊκό Εμπορικό Κώδικα. Πριν όμως ε, έχουμε στη διάθεσή μας ένα τέτοιο κώδικα, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση, να θέσω μια ερώτηση πιο πραγματιστική, αν θέλετε. Για το κοινό πλαίσιο αναφοράς, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρξουν αλλαγές και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας και το χρονοδιάγραμμά σας για τις μεθόδους οι οποίες προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων που έχετε ε, σε επίπεδο του δικαίου συμβάσεων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης με τη νέα μου γενική διεύθυνση βρήκα αυτό τον τόμο του κοινού πλαισίου αναφοράς. Ξέρω ότι εσείς έχετε δουλέψει πάρα πολύ σαν βουλευτές γύρω από αυτό το, το, το, το, κώδικα και θέλω να προχωρήσω γρήγορα. Θέλω να προχωρήσω γρήγορα γιατί πρέπει ο κώδικας αυτός, το βιβλίο αυτό αν θέλετε, να μην γίνει μόνο αντικείμενο πανεπιστημιακής χρήσης και μελέτης, αλλά να τεθεί πλήρως σε ισχύ και σε εφαρμογή. Και έτσι λοιπόν ήδη κατά τη διάρκεια του 2010 θα επεξεργαστούμε την ουσία του CFR, του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς, και ελπίζουμε ότι ήδη το καλοκαίρι του 2010 αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα ασχοληθεί θα εκδώσει μία ανακοίνωση. Και το 2011 ελπίζω να έχουμε συγκεκριμένο νομικό μέσο για χρήση. Γνωρίζω ότι ήδη οι πανεπιστημιακοί έχουν ξεκινήσει τις μεταφράσεις γιατί το CFR, το κοινό πλαίσιο αναφοράς, είναι στα αγγλικά. Έχουν προχωρήσει οι γαλλικές και γερμανικές μεταφράσεις και θα ήθελα να συνεχιστεί η προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να βοηθήσει για να ολοκληρωθεί η δουλειά αυτή. Συμπληρωματική ερώτηση. Μιλήσατε για τους πανεπιστημιακούς, πώς ε, θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει στην εφαρμογή του CFR. Επαναλαμβάνω ότι η ανακοίνωση το καλοκαίρι του 2010 θα δώσει τη δυνατότητα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει απόλυτα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην διάθεσή του και να δει αυτό τι θέλει να κάνει από εκεί και πέρα. Και γι' αυτό θα ξεκινήσει ε, με την ανακοίνωση η διαδικασία και όχι με μία πρόταση για απόφαση γιατί θεωρώ πάντα σχεδόν ότι πριν φτάσει κανείς σε συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να προσπαθήσει να συγκεντρώσει την πλήρη σοφία όχι μόνο των ακαδημαϊκών πανεπιστημιακών αλλά και αυτών οι οποίοι σε καθημερινή πρακτική βάση ασχολούνται με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, δικηγόροι, δικαστικοί, εισαγγελείς και πολιτικοί φυσικά και με βάση ακριβώς αυτή την κοινή θα έλεγα σοφία, την κοινή με την έννοια την διαθέσιμη σε όλους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε προτάσεις νομικών μέσων. Ε, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μια συζήτηση ευρεία γύρω από το CFR και αυτό δεν ήταν σωστό. Όπως είπα, εγώ δεν είμαι ειδική σε, σε τέτοια θέματα και θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Θέλω να καταλήξει θετικά η διαδικασία αυτή γιατί είναι πράγματι το έμβριο αν θέλετε που κάποια στιγμή θα οριμάσει και θα οδηγήσει στον Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα, λέει η κυρία Λίχτενμπέργκερ, που αφορά άμεσα την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι στην εφαρμογή του, εθνικού, του κοινοτικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες και πάρα πολλά παράπονα από τους συμπολίτε ε, και έχουμε όμως ταυτόχρονα και λιγότερες διαδικασίες επί παραβάση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ιδιαίτερα στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Ε, γίνεται τα τελευταίο καιρό λιγότερα πράγματα από ό,τι παλιότερα Πώς ακριβώς λοιπόν θα προχωρήσουμε, πώς ε, θα ελέγχεται η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ξέρετε ότι θα υπάρξει σύντομα μια νέα διοργανική συμφωνία. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής δεν θα έπρεπε να υπάρξουν πρακτικά μέτρα για τη συνεργασία του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο συγκεκριμένο τομέα. Μήπως θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει και να ελέγχει και αυτή με τη σειρά της κάποιες τέτοιες διαδικασίες μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου. Έχετε απόλυτα δίκιο όταν λέτε ότι δεν αρκεί κανείς το ευρωπαϊκός νόμος όταν ο νόμος αυτός μόνο εν μέρη ή και καθόλου δεν περνά σε ε, εθνικό νόμο και δεν γίνεται ε, θεμελιώδες δικαίωμα. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σαν Επίτροπος Αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες είχα χρησιμοποιήσει όχι την οδηγία αλλά τον κανονισμό σαν μέσο γιατί ο κανονισμός ήταν και πιο ταχύς και de jure επέτρεπε την εφαρμογή του άμεσα. Τώρα εδώ βρίσκομαι σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα, βέβαια έναν τομέα πάρα πολύ ευαίσθητο και έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο ποινικό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κανονισμούς. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο αστικό. Έχω πράγματι υποσχεθεί εφόσον θα μου το επιτρέψετε να έρχομαι μπροστά σας μία φορά κατέτος με μία έκθεση για την εφαρμογή ε, των θεμάτων των θεμελιωδών ελευθεριών και ε, δικαιωμάτων και σε επίπεδο ευρωπαϊκού νόμου αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχει κατέτος μια συλλογή όλων των παραπώνων που φτάνουν σε εμά και από την Επιτροπή Αναφορών, από όλους εσάς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον διαμεσολαβητή, τον Ombudsman και όλα αυτά να αναλύονται αφού συλλεγούν για να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός. Και θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ δεν θα διστάσω να ξεκινήσω διαδικασίες επί παραλήψη. Αν δείτε το τι έχω κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια θα κατανοήσετε ότι δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπερβολικά φοβισμένη να λέω τη γνώμη μου ακόμα και στις μεγάλες χώρες μέλη. Ιδιαίτερα ικανοποιητική η απάντησή σας, έτσι ε, αυτή είναι η πρώτη μου εντύπωση, αλλά αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον όταν ε, θα υπάρχει το follow-up σε θέματα που θα έχουν σχέση με τις εκθέσεις για το κοινοτικό δίκαιο, εκθέσεις που υποβάλλονται από ευρωβουλευτές, μπορώ να θεωρήσω ότι τότε θα μας δίνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί αυτό δεν συνέβη τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το εξασφαλίσουμε γιατί σε τελική ανάλυση εδώ ε, έχουμε κοινοβουλευτικά καθήκοντα και βεβαίως και η Κομισιόν έχει κάποια καθήκοντα ως θεματοφύλακας του κοινοτικού δικαίου. Τις ε, τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος κύριος Μπαρόζο ε, κάλεσε επανειλημμένα τους υποψήφιους επιτρόπους ε, να συζητήσουν ακριβώς για αυτά τα θέματα. Κατέστησε λοιπόν απόλυτα σαφές ότι αυτός ο ακόμα πιο σημαντικός ρόλος του Κοινοβουλίου τώρα πλέον ε, βάσει της ε, συνθήκης. Αυτός ο ρόλος απαιτεί άμεσες ε, απαντήσεις εκ μέρους των ε, Επιτρόπων προς το Κοινοβούλιο. Τώρα εγώ το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι το τι θα κάνω εγώ. Τα τελευταία δέκα χρόνια και μπορείτε να ρωτήσετε τις επιτροπές που συνεργάστηκα μαζί μου, ήμουνα πάντα παρούσα οποτεδήποτε το Κοινοβούλιο θέλησε να συζητήσει μαζί μου. Και εξάλλου και εγώ ζήτησα από το Κοινοβούλιο να συζητήσουμε οποτεδήποτε έκρινα ότι χρειαζόμουν την άποψη του Κοινοβουλίου. Και τα κοινοβουλευτικά θέματα βεβαίως πρέπει να απαντώνται ταχύτατα γιατί εσείς είσαστε ο διάμεσος κρίκος ε, που μας συνδέει με τους Ευρωπαίους πολίτες. Επόμενος συνάδελφος. Κάριμ. Από τη μια μεριά λέτε ότι δεν σας αρέσει να μην προχωράει ενιαία μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα μπρος. Από την άλλη μεριά δεν έχετε ικανοποιητικέ απαντήσεις όταν σας ρωτάμε για την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τον τρόπο με τον οποίο δρά. Μερικές φορές αναγκάζει τις χώρες οι οποίες ακολουθούν το κοινοτικό δίκαιο να αποκλείονται από συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους. Γι' αυτό το θέμα δεν έχετε καμία απάντηση. Μιλάτε για τη συνθήκη της Λισαβόνας που προβλέπει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με σεβασμό των διαφόρων νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών. Εσείς στην γραπτή σας απάντηση στο ερωτηματολόγιο που σας δώσαμε και σε αυτά που μας είπατε στην αρχή, είπατε ότι η πρόθεσή σας είναι να περάσετε από το πρώτο κομμάτι συμβατικού δικαίου στο αστικό. Εσείς με ένα αστικό δικαστήριο τι θα κάνετε, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παραδόσεις των χωρών ε, μελών και το εθνικό δίκαιο. Είναι πολύ σημαντικό να προωθείτε αυτό το δίκαιο. Έχω και διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την τρέχουσα ε, πρόταση για την διαθήκη, τα κληρονομικά δικαιώματα κλπ. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης δεν προβλέπει ε, ομοιομορφία στο συμβατικό δίκαιο. Εσείς θα πάτε ακόμα πιο πέρα και αν ναι, με ποια εντολή, από πού σας έχει έρθει μια τέτοια εντολή για να το κάνετε. Το μόνο που μπορώ να απαντήσω, λέει κύριε Ρέντινγκ, είναι αυτό το οποίο απάντησα και στην αντιπρόεδρο Wallis πριν για το ίδιο αυτό θέμα. Ότι δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση και για τους 27. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο όσον αφορά το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα κάνω ανακοίνωση αφού προηγουμένως έχω ακούσει τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν και εμπειρογνώμονες ε, του κοινού δικαίου. Όμως, τελικά, στο τέλος, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία λύση. Ή εντάξει, ας μην πω λύση, ας πω πρόταση, γιατί εγώ πρόταση θα σας υποβάλω για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, ώστε τα δικαιώματα των πολιτών, εάν πάνε στο εξωτερικό, να λαμβάνονται ακόμα υπόψη. Τώρα για το πιο ειδικό θέμα όσον αφορά τις διαθήκες. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει ένα ειδικό στοιχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχει ληφθεί υπόψη το στοιχείο αυτό στο έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου αυτή η ιδιαιτερότητα που αφορά τους Βρετανούς που ζουν στο εξωτερικό να ληφθεί υπόψη. Και αν δεν με πατάει μνήμη μου, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη, 95% σίγουρη είμαι, μπορούν να επιλέξουν οι Βρετανοί αν θέλουν να εφαρμοστεί το Βρετανικό σύστημα ή αν θέλουν να εφαρμοστεί το σύστημα του κράτους μέλους κατοικίας τους. Η δουλειά συνεχίζεται για αυτό το θέμα πάντως. Συμπληρωματική ερώτηση. Εσείς αναφέρεστε σε προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ακριβώ επειδή δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τον, τη χώρα διαμονής και κατοικίας. Όμως, για αυτά που μας είπατε κύριε Επιτροπέ και όσον αφορά το μέλλον ε, και σχετικές νομοθετικές ε, προτάσεις εσείς θα στηρίξετε την αξιολόγηση από πλευρά των κρατών μελών. Εγώ δεν ξέρω τι εννοείται με την αξιολόγηση αυτή στα κράτη-μέλη. Εμείς πάντα έχουμε δύο αξιολογήσεις αντικτύπου. Η μία λαμβάνει υπόψη το κάθε ένα σύστημα από τις 27 χώρες μέλη, αν αυτό εννοείται, τότε η απάντησή μου είναι ναι. Και έχουμε και επιπλέον αξιολόγηση αντικτύπου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διπλή αξιολόγηση, διτή. Αυτό το δεύτερο προστίθεται τώρα, δεν υπήρχε πιο πριν. Υπάρχουν και θεμελιώδη δικαιώματα και για την ελεύθερη κυκλοφορία. Και αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχουμε επιτέλους σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε και το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νομική ευρωπαϊκή τάξη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουν, να συνειδητοποιούν τα δικαιώματά τους οι Ευρωπαίοι πολίτες και τις δυνατότητες πρόσβασης στο σύστημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η νομική νοοτροπία επίσης των εθνικών χρηστών του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή δικηγόρων και δικαστών που είναι οι πρωταγωνιστές στον τομέα αυτό. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να συνεχίσετε να προετοιμάζετε σωστά τους Ευρωπαίους, τι περισσότερες επενδύσεις θα κάνετε, πώς θα ε, στηρίξετε τα network, τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν και τις επιμορφωτικές διαδικασίες και πώς θα ενισχύσετε τις διαδικασίες αυτές σε εθνικό επίπεδο. Πώς ε, θα μπορέσετε να εμπλέξετε ε, και τα πανεπιστήμια στα πλαίσια ενός συστήματος το οποίο να προπαρασκευάζει ακριβώς τους πρωταγωνιστές του νομικού συστήματος για να οδηγηθούμε στην αμοιβαία αναγνώριση και τον αμοιβαίο σεβασμό των διαφορετικών νομικών διαδικασιών. Έχετε απολύτως δίκιο. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορεί με διάταγμα να επιβληθεί εκ των άνω. Υπάρχει γιατί οι χρίστες χρήστες της γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε μία χώρα, το τι συμβαίνει στην άλλη χώρα και γνωρίζουν την αντικειμενική σοβαρότητα με την οποία και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο όταν ήμουν επίτροπος για την παιδεία επέμενα για την βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος Εράσμους έτσι ώστε και τα πανεπιστήμια να μπορούν να παρέχουν ένα κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισότιμο δίπλωμα μάστερ. Ακριβώς γιατί οι νέοι οι οποίοι σπουδάζουν σε διάφορα πανεπιστήμια και σπουδάζουν με καθηγητές διαφορετικών νοοτροπιών και πρακτικών, όταν επιστρέφουν στην χώρα τους να μην έχουν νομικά προβλήματα και να μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρη ευρωπαϊκή λογική. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα πετύχουμε ε, δημιουργία ενός εράσμους για δικαστές. Δικαστές από τη μια χώρα που να αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα των νομικών συστημάτων των υπολείπων χωρών. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε μια ουσιαστική αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της νομικής σκηνής. Φυσικά και πρέπει να ενισχύσουμε τα υπάρχοντα δίκτυα, υπάρχει το φόρουμ για τη δικαιοσύνη, πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε περιλήψεις των νομολογιών, να βοηθήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση, και εγώ εκεί σίγουρα θα χρησιμοποιήσω τα πολύ καλά Ινστιτούτα και νομικά πανεπιστήμια που έχουμε σε όλη την Ευρώπη και θα προσπαθήσω όλα αυτά να τα συνδυάσω, να τα καταστήσω διαλειτουργικά. Και στο τέλος, ποιος ξέρει, ίσως, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, αλλά αυτό σε επίπεδο δικτύου σε μια πρώτη φάση. Ευχαριστώ Επίτροπε. Υπάρχει ένα είδος εράσμος για τους δικαστές, αλλά αφορά μόνο έναν στους χιλίους, ένα πολύ χαμηλό αριθμό δηλαδή. Και γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία διεξάγεται και υπάρχει στις διάφορες ε, χώρες ε, βασίζεται στα μαθήματα εκ των άνω σαν να μαθαίνει κανείς πράγματα στον πρόεδρο του δικαστηρίου θεωρώντας ότι είναι μαθητής ένας πρόεδρος δικαστηρίου. Μήπως θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων επαγγελμάτων και κυρίως των νομομαθών βασιζόμενοι στις πρακτικές και στις, ε, στις μεθόδους που χρησιμοποιούν στα δικά τους συστήματα. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της κατάρτισης των ενηλίκων πάντα βέβαια. Αυτό θα ήταν ε, πράγματι ο στόχος μιας τέτοιας Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Δικαίου, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, ό,τι και να κάνουμε εμείς Ακόμα και αν έχουμε ένα εκατομμύριο φοιτητέ Εράσμου, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών δεν είναι παρά μία σταγόν εν το ωκεανό. Συνεπώ θα πρέπει όλα αυτά μένα να τα ενισχύσουμε, αλλά να ενισχύσουμε εμείς επίσης και τις πρακτικές πλευρές, χωρίς να ξεχνάμε την ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή έρευνα. Ξέρω σαν παράδειγμα τι γίνεται στην χώρα σας, στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, όπου θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Ιταλία γύρω από την έρευνα στον τομέα το νομικό και επίσης ε, να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες ε, που ε, προσφέρει η διαδικασία αυτή και στους Βρετανούς συναδέλφους που έχουν ανησυχίες σχετικά με τη νομική τους παράδοση. Κυρία Ρέντινγκ, Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, παρουσίαση της εργασίας μας ε, προς ε, την κοινή γνώμη προς τα έξω. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας υποβάλω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά σε θέματα δικαίου. Ως μέλος της Επιτροπής της Νομικής έχω διαπιστώσει επανειλημμένα ότι στα μέσα ενημέρωσης προβάλλονται τελείως διαφορετικά θέματα από αυτά που εξετάζονται στη δική μας την Επιτροπή τη Νομική. Στο δικό σας το χαρτοφυλάκιο θα υπάρξουν θέματα όπως ε, το σκάνερ ε, σώματος και με βάση τις ε, ερωτήσεις που μας δώσετε σε γραπτή μορφή, εσείς θα ασχοληθείτε πρώτα απ' όλα με θέματα οικογενειακού δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ πολύ συγκεκριμένα. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς επιδιώκετε στο θέμα του οικογενειακού δικαίου πέρα από το ΡΟΜΗ 3 και ως πρώην δημοσιογράφος τη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Πώς ακριβώς προτίθεστε να την προβάλλετε περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου στον τομέα αυτό, αναφερθήκατε σε αυτήν, ε, είναι φρικτό και για μένα. Ε, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ε, εγώ γεννήθηκα δημοσιογράφος ε, και εξακολουθώ να αισθάνομαι δημοσιογράφος. Δεν μπορεί κανείς να γράψει μια καλή ιστορία αν δεν υπάρχει καπνός. Χρειάζεται δηλαδή κανείς ένα γεγονός για να γράψει μια καλή φωτιά, μια καλή ιστορία. Και όσον αφορά το κοινό πλαίσιο αναφορά, ίσω ε, να μην μπορέσουμε να τραβήξουμε την προσοχή των μέσων ενημέρωση. Συγγνώμη, Λένα. Αλλά για τα οικογενειακά, παρήματο χάρη. Αν ξεκινήσουμε από τα συγκεκριμένα ε, παραδείγματα από άτομα, αν αναφέρουμε συγκεκριμένα, ε, τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτό που σα είπα, το παράδειγμα Μικτού γάμου τι πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι αν ένας ε, Φινλανδός ε, θέλει να παντρευτεί μια Βρετανίδα αλλά όπως σας είπα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται δεν υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση ή αυτές οι φρικτές ιστορίες της ε, απαγωγής παιδιών ή του αδύναμου κρίκου σε ένα γάμο που υφίσταται τα πάντινα λόγω της απόφασης του δικαστηρίου. Για όλα αυτά πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να τα προβάλλουμε προς τα έξω. Ξεκινώντας με το πρόβλημα του πολίτη και το πώς λύνουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ε, Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν. Βλέπω ότι σιγά, σιγά έρχονται μέσα στην αίθουσα και τα μέλη της Επιτροπής ε, Γυναικών. Ας πάμε στο θέμα της ε, βίας έναντι των γυναικών. Ποιες είναι οι δράσεις που θα αναπτύξουμε, με βάση ποιο πρόβλημα. Να εντάξει, να το εξηγήσουμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Το Κοινοβούλιο κάνει κάτι συγκεκριμένο για τους πολίτες. Αυτές είναι οι ιστορίες που περνάνε στην κοινή γνώμη. Και εμείς πρέπει να ε, συστήσουμε την βάση, την ουσία των ιστοριών για να περάσουν και οι ιστορία μας, ιστορίες μας στα μέσα ενημέρωση. Και συμπληρωματική ερώτηση. Ελπίζω ότι η, δική μας, ε, η δουλειά της δική μας Επιτροπής θα είναι σε καλά χέρια σε εσά και να μην είμαστε ουραγοί πίσω από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Με τον ε, κύριο Μπαρόζο θα ξεκολουθείτε να είσαστε αρμόδιοι για την επικοινωνία και ε, με όλα αυτά ε, πώς μπορεί να ε, διαφυλαχθεί η ουδετερότητα που, των επιτρόπων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ο διαχωρισμός σε τελική ανάλυση του δικού σας του χαρτοφυλακίου με άλλα γενικότερα θέματα ο διαχωρισμός πώς μπορεί να γίνει χωρίς βέβαια να υποστεί ζημιά το δικό σας το χαρτοφυλάκιο. Θα πρέπει την επικοινωνία να την προβάλλω πολύ πιο συγκεκριμένα. Όλοι σας εδώ στην αίθουσα έχετε μεγάλη εμπειρία και πολλοί από εσάς ε, έχετε συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές εκλογές. και είδατε πράγματα που ε, τα βίωσαν όλοι οι πολίτες, γιατί τα βίωσαν στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι λοιπόν εμείς, και όταν λέω εμείς ενώ και εσάς ως ε, μέλη του Κοινοβουλίου, κάθε ε, μεμονωμένος ε, βουλευτής έχει να πει μια δική του συγκεκριμένη ιστορία. Αυτές λοιπόν τις ιστορίες θα προβάλλουμε και θα τις εξηγήσουμε στους πολίτες. Έχουμε λοιπόν επικοινωνία η επικοινωνία ενημέρωση ε, που έχει άμεση σχέση με συγκεκριμένες δράσεις. Πρέπει ε, να εξηγήσουμε στον πολίτη βεβαίω και πράγματα πολύ πιο γενικά, οριζόντια, το τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτόν και αυτό αφορά τόσο την ελεύθερη μετακίνηση όσο και τα κοινωνική φύσεω και περιβαλλοντικής φύσεως θέματα. Ο κάθε επίτροπος έχει να πει τα δικά του ε, και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών ε, θα έχει ως στόχο να συγκεντρώνει όλες αυτές τις απόψει για να γίνονται κατανοητές από ε, τους Ευρωπαίου πολίτες. Αντώνιο Λόπες Βάιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ αναγνωρίζουμε την μακρά σας εμπειρία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εσείς γνωρίζετε τις ανησυχίες της Επιτροπής μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εσωτερική αγορά οι πολίτες. Ξέρετε και τις επιτυχίες της Επιτροπής μας να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 125 της Συνθήκης. Δεν υπήρξαν πολλέ δράσει από την Κομισιόν κατά το παρελθόν. Τώρα έχουμε το δημογραφικό ζήτημα, τη γύραση του πληθυσμού τι συγκεκριμένη δράση σκοπεύετε να αναλάβετε μετά από την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ευάλωτους ενήλικες και προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να βελτιωθεί η αναγνώριση αποφάσεων για την προστασία ενηλίκων όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Ε, θα έχουμε όλο και περισσότερους ευάλωτους ενήλικες, δεδομένου ότι γερνάει η κοινωνία μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όταν μιλάμε για διακρίσεις και για την οδηγία για τις διακρίσεις, σπάνια μιλάμε για την γύρανση του πληθυσμού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πραγματικά οριζόντιο ζήτημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Στο τρέχον σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα κενό για την περίπτωση αυτή των ευάλωτων ατόμων, των ηλικιωμένων ατόμων που έχουν ε, αναπηρίες ε, είτε σωματικές είτε διανοητικές. Υπήρξε σύμβαση του 2000 και είναι μια καλή αρχή. Ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή. Όμως, τίθεται σε εφαρμογή σε ορισμένες μόνο χώρες μέλη. Και πιστεύω ότι θα μπορούσε να διευκρινιστεί περισσότερο μέσω μιας κοινοτική νομοθεσίας, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τώρα, αυτή η νομοθεσία πώς θα πρέπει ακριβώς να έχει, μένει να το δούμε. Αλλά και εδώ πάλι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα ήθελα να βοηθήσετε κι εσείς. Και θα ξεκινήσω μία μελέτη αξιολόγησης για να δω ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα και ε, τι μεταχείριση έχουν στις διάφορες χώρες. Αν υπάρχουν καλές πρακτικές, να τις χρησιμοποιήσουμε. Ούτε αποκλείω βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, δεν αποκλείω ούτε και μια νομοθετική πρόταση. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μετά την μελέτη αξιολόγησης και μετά τις συζητήσεις που σκοπεύω να έχω με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε πει αυτό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα γίνει ακόμα πιο σοβαρό μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε. Συμπληρωματική ερώτηση δεν έχετε, οπότε επόμενος ο κύριος Έγκστρομ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μ' άρεσε η απάντηση που δώσατε στην κυρία Ρουγκεν νωρίτερα. Είπατε ότι θέλετε να προχωρήσετε με μια πρωτοβουλία όσον αφορά τα πλαστά προϊόντα αλλά δεν μιλήσατε για κυρώσεις και κατά τη γνώμη μου είπατε κι εσείς ότι το downloading τελείως διαφορετικό από τα πλαστά προϊόντα είναι όντω διακριτές περιπτώσεις. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε θα αντικαταστήσει την οδηγία περδίο που συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω αυτά τα γεγονότα. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να ρωτήσω τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή να μου εξηγήσει περισσότερο. Είναι μια οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε. Το δεύτερο όμως για τις κυρώσεις, όχι. Πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται. Η κυρία Ρέντινγκ, εγώ μιλούσα για ποινικά ζητήματα όσον αφορά τα πλαστά προϊόντα. Η πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβουμε από κοινού με την Σεσίλια Μάλστρομ, διότι εκείνη είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της απάτης. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε. Αλλά για την πρόσβαση τώρα στο διαδίκτυο και το copyright εδώ δεν πρόκειται για το ίδιο. Δεν πρόκειται για πλαστά προϊόντα εδώ, για παραπίση Είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς επειδή είχαμε μια μεγάλη συζήτηση, μάθαμε πολλά. Και το ξέρετε κι εσείς ότι η συζήτηση δεν έγινε μόνο εδώ σε αυτό το σώμα, έγινε και στα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται συνειδητοποίηση Καταρχήν, για να προστατεύσουμε την δημιουργία στο διαδίκτυο. Και η συνειδητοποίηση αυτή υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να ενισχυθεί, να προστατευτεί η πραγματική δημιουργία με τα μέσα που είχαμε παλιά στη διάθεσή μας. Χρειάζονται νέα μέσα, διασυνοριακά. Εγώ έχω θέσει επιτάπητος και έχω προτείνει κάτι μαζί με τον συνάδελφο Μακρύβη για το copyright online στο διαδίκτυο. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να χειριστούμε το θέμα αυτό του copyright στο διαδίκτυο. Υπάρχει και ο συνάδελφος Μισελ Μπαρνιέ και ο συνάδελφος Νέλη Κρούς και όλοι μαζί πρέπει να φροντίσουμε να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εφόσον επιθυμείτε και επιβεβαιώσετε τον ορισμό μου στη θέση της Επιτρόπου, τότε θα φροντίσω και για τα θεμελιώδη δικαιώματα οριζοντίως να τεθούν σε εφαρμογή και σε αυτή την πρόταση που ελπίζω ότι θα βγει με τη συνεργασία μας. Γιατί πιστεύω και εγώ ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες, κάθε μία και όλες τις αποφάσεις που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασε το χρόνο μου, να σταματάω. Ε, συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Έξτρομ. Όχι, εντάξει ικανοποιήθηκα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, τελευταία ερώτηση. Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω. Είπα ήδη και προηγουμένως ότι ε, είναι θέμα συζήτησης σε διάφορα θέματα. Θέμα συζήτηση για διάφορα θέματα. Υπάρχουν δηλαδή θεμελιώδη δικαιώματα που δεν μπορεί κανείς να τα διχοτομήσει ή ε, άλλα που δεν μπορούν να συζητηθούν. Παραδείγματο χάρη, η θανατική ποινή. Αυτή δεν μπορεί να επανέλθει. Τελεία. Αλλά υπάρχει παραδείγματο χάρη το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία. Υπάρχει το δικαίωμα δίκαιης αποζημίωσης, το δικαίωμα του copyright. Ε, πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσει κανείς ε, τα διάφορα ε, δικαιώματα που θα μπορούσαν να συγκρουστούν και να βρει κάποια λύση. Νομίζω λοιπόν το θέμα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο και για την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να διεξάγουμε σοβαρά σοβαρέ Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία τώρα ερώτηση. Από τον κύριο Τσιόμπρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Όμως ε, Όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση, είχαμε, σημειώσαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά πρόκειψαν και κάποιοι κίνδυνοι καθοδόν. Τι εννοώ? Υπάρχει ο κίνδυνος ελεύθερης μετακίνησης ε, ε, εγκληματιών εις βάρος των παιδιών που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος των παιδιών. Μήπως λοιπόν προτίθεστε να συντάξετε ε, έναν κατάλογο, ένα μητρό αυτών των ανθρώπων που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών. Και μία άλλη ερώτηση. Όλοι μας ε, πιστεύουμε ότι η κατάσχεση ε, περιουσιακών στοιχείων είναι ε, μία πολύ αποτελεσματική μέθοδος κατά της μαφίας. Πιστεύετε εσείς ότι μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε όσον αφορά τέτοιου είδου ενέργειες, να επιβάλλεται δηλαδή κατά σχέσεις σε ορισμένε χώρες. Γιατί υπάρχουν κάποια τέτοιου είδου μέτρα που εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και σε άλλες ή ενδεχομένω και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι η παιδοφιλία είναι ένα ιδεχθέστατο έγκλημα και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ε, εξαφανιστούν από προσαπογείς οι παιδεραστές. Και σίγουρα να μην μπορούν αυτοί να ε, εργάζονται διασυνοριακά. Γιατί πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ένα διασυνοριακό έγκλημα η συνάδελφός μου, κυρία Σεσίλια Μάλστρομ και εγώ θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε απόλυτα συγκεκριμένα για να βοηθήσουμε την αστυνομία να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα ε, στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών για να εξαλειφθεί όπως σας είπα αυτή η απαράδεκτη στάση ζωής. Τώρα, όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την ανάσχεση του οργανωμένου εγκλήματος, εδώ περνάμε στον τομέα του ποινικού δικαίου. Και όπως επανειλημμένα έχω πει, στο ποινικό δίκαιο η αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων, η συνεργασία, η διασυνοριακή πρέπει πράγματι να ισχύει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στις προτάσεις που καταθέτουμε γιατί ε, πάντα υπησέρχεται το στοιχείο της επικουρικότητας. Πρέπει λοιπόν να συμπεριλαμβάνονται και τα εθνικά κοινοβούλια και αν καταθέσουμε μια σχετική πρόταση ε, μπορεί ενδεχομένως ε, μια κυβέρνηση να μας μπλοκάρει βασιζόμενη στο επιχείρημα sui generis. Εγώ θεωρώ ότι εγκλήματα που δεν συζητούνται είναι, όπως σας τα είπα, οι δεχθέστατα. Και η παιδεραστία για μένα κατατάσσεται σε αυτά. Πρέπει λοιπόν να ε, βρούμε τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουμε. Όταν εγώ ήμουνα επίτροπος για τις ε, τηλεπικοινωνίες, συνεργάστηκα με βιομηχανικούς κύκλους. Χτυπάει το καμπανάκι και ε, δεν τελειώνει καν τη φράση της η κυρία Επίτροπος. Διακόπτεται. Ε, πρόεδρος, ε, λυπάμαι που σας ε, διάκοψα, αλλά πρέπει να είμαστε σύντομοι για να σεβαστούμε και την Επιτροπή Γυναικών. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, ολοκληρώστε. Συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, ε, όσον αφορά αυτά που μας είπε η κυρία Επίτροπος, Θέλω να μας πείτε για την εμπειρία σας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι μπορούν να γίνουν ε, πολλά περισσότερα όσον αφορά την ε, διαβίβαση δεδομένων Αναφέρομαι κυρίως σε, σε πληροφορίες για εγκληματίες, για παιδεραστές. Ε, ξέρω ότι τέτοιου είδους ε, πληροφορίες μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες ε, για να προστατευθούν παιδιά από παιδεραστές. Κοιτάξτε, αυτό που έκανα τότε που ήμουν επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες ήταν κυρίως να βελτιώσω, να ενισχύσω τη συνειδητοποίηση του θέματος. υπήρχε ένα πρόγραμμα στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των εκπαιδευτών, των γονέων, γιατί δεν μπορεί κανείς ε, να εμποδίσει τα παιδιά στο να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Όμως μπορεί κανείς να τα ενημερώσει για τους κινδύνους. Συνεργασία λοιπόν με την, ε, τους αρμόνιους, ε, αρμόδιους βιομηχανικούς κύκλους. Συμφωνήσαμε κάποιες μορφές επικοινωνίας να τις ε, απομακρύνουμε από τα κινητά τηλέφωνα της ε, τρίτης γενιάς. Και κοινωνικά δίκτυα επίσης. 21 βιομηχανικοί κλάδοι υπέγραψαν μία συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2010 όταν θα συζητηθεί το προφίλ του ανήλικου. Να μην είναι εύκολο να τον πλησιάσει κανείς. Μπορώ λοιπόν να σε αναφέρω μια ολόκληρη σειρά μέτρων ποινικοποίηση αλλά και μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται τα παιδιά όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε ε, και τώρα για να ε, προχωρήσουμε γρήγορα δίνω ε, το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών και μία επισήμανση θα μου επιτρέψετε η συνεδρίαση των συντονιστών ε, της Επιτροπής της Νομικής είναι στις 4.30 και ε, στις 5 ε, η ώρα θα ακολουθήσει η κανονική συνεδρίαση των, της, της Νομικής Επιτροπής. 4.30 οι συντονιστές και 5 η Νομική Επιτροπή. Συνεχίζουμε με την ακρόαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ίσων Ευκαιριών. Θα ακολουθήσουμε την ίδια αρχή, όπως έγινε και με τους συναδέρφους στις προηγούμενες επιτροπές. Έχουμε στη διάθεσή μας μισή ώρα Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Μπορώ να σας πω όμως ήδη ευθύ εξ αρχής ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Ένα λεπτό για τις ερωτήσεις, δύο λεπτά για κάθε απάντηση. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο βέβαια στην κυρία Ρέντινγκ. Για τρία λεπτά παρακαλώ κυρία Ρέντινγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Έχω μόνο 30 λεπτά στη διάθεσή μου. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι πολύ σύντομη στην εισαγωγή μου, να που έχουμε μόνο 30 λεπτά για να συζητήσουμε, για να περάσουμε μετά στις ερωτήσεις σας. Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ με την Επιτροπή Γυναικών, διότι ο κύκλος έκλεισε, θα έλεγα. Βλέπετε, ξεκίνησα την πολιτική μου ζωή ως συγγήτρια στο Εθνικό Κοινοβούλιο της ε, χώρας μου υποβάλλοντας οδηγία ε, για νόμο όσον αφορά την ίση μεταχείριση. Έπειτα πήγα και πρόεδρος των ε, ε των χριστιανοκοινωνικών συγγνώμη, γυναικών στο Πεκίνο για να εκπροσωπήσω τις γυναίκες εκεί. Και εδώ χαίρομαι λοιπόν γιατί βρίσκομαι μπροστά σε ένα σωρό γνωστά πρόσωπα. Θα είμαι σύμμαχός σα κάθε φορά που θέλουμε να ενισχύσουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σε κάθε τομέα της πολιτικής μας. Και μπορείτε να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μειώσω το χάσμα που υπάρχει όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο πρόεδρος Μπαρόζο θέλησε να μου αναθέσει και την αρμοδιότητα των οδηγιών και την καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με το ποινικό δίκαιο. Όπως επίσης θέλησε να μου αναθέσει και τους μηχανισμούς για να καταπολεμηθεί η βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου για να πετύχουμε μια πραγματικά ισχυρή και με προβολή πολιτική όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σκοπεύω επίσης και τις δραστηριότητε επικοινωνίας να τις ε, βάλω στην υπηρεσία της δουλειά μου αυτής. Θέλω να χρησιμοποιήσω κάθε δυνατότητα, κάθε μέσο, κάθε μηχανισμό που έχω στη διάθεσή μου για να φροντίσω να είμαι πραγματικά η Επίτροπος Ισότητας των δύο φύλων. Το μέτρο θα είναι πάντα και ο γνώμονας η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι τώρα πια είναι δεσμευτικός και ότι έχουμε και το άρθρο 23 ε, του χάρτη αυτού που διασφαλίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς και στην απασχόληση και στην πληρωμή. Και ακριβώ επειδή έχω την οριζόντια ευθύνη να θέσω σε εφαρμογή τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς σε όλες τις αρμοδιότητες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κοιτάξω αν κάτι δεν πάει καλά με την ισότητα των φίλων να παρέμβω. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις σας τώρα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ρέντινγκ, θα ξεκινήσω λοιπόν με την κυρία Μπάουερ. Παρακαλώ κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Προτινόμενη Επίτροπε, Φυσικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που ακούμε από εσά, ότι δηλαδή δεσμεύεστε υπέρ τη ισότητα των δύο φύλων. Σε αυτό το θέμα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κοινοτική νομοθεσία, πολύ κοινοτική νομοθεσία και κάθε αλλαγή κοστίζει πολύ σε χρόνο. Ανάμεσα στο Γιούρι και την de facto ισότητα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αν δούμε όλο το πακέτο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στην πληρωμή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και τελευταία, οι οικονομολόγοι λένε ότι οι διαφορές Αυτέ, στου μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν και άμα μια γυναίκα αφήσει τη δουλειά τη για μερικά χρόνια για να κάνει παιδιά και να ασχοληθεί μαζί του και μετά επιστρέψει στην αγορά εργασία. Τι άλλο εκτό από διάκριση είναι αυτό. Θέλω λοιπόν μια απάντηση από εσά. Τι σκοπεύετε να κάνετε πρώτα απ' όλα για να τελειώσει αυτή η διάκριση. Διότι εμεί δεν θέλουμε να έχουμε διατάξεις που να παραμένουν νεκρό γράμμα του νόμου Ευχαριστούμε. Κυρία Ρέντι. Ευχαριστώ. Ε, έχετε απόλυτα δίκιο. Παρά όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, εξακολουθούν να παραμένουν διαφορές της τάξης του 17%. Πράγματι. Είναι απαράδεκτο. Και γι' αυτό και ο αγώνας κατά της διαφοράς αυτής τους μισθούς θα αποτελέσει και μία από τις προτεραιότητές μου. Μάλιστα αναφέρεται και ρητά στη συνθήκη, πρέπει να ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι έχουμε παραπάνω δυνατότητες για νομοθετική και μη νομοθετική δράση και μέτρα σε αυτό το τομέα. Φυσικά και πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να οδηγηθούμε σε λύσεις. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέσο στη διάθεσή μας που εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά μέχρι τώρα. Κάθε άνοιξη έχουμε ε, μια στρατηγική για την απασχόληση. Δεν θα ήθελα σε αυτήν την στρατηγική κάθε χρόνο να προστίθεται ένα χαρτί για την ισότητα των φύλων. Όχι, θέλω η ισότητα των φύλων να εφαρμοστεί πλήρως στην στρατηγική αυτή για την απασχόληση. Χαίρομαι πάντως που η Βελγική Προεδρία έχει ήδη πει ότι η κάλυψη της διαφοράς αυτής θα αποτελέσει προτεραιότητα της Προεδρίας της. Θα επικεντρωθούν σε αυτό δηλαδή στη Βελγική Προεδρία. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε με όλες τις δράσεις που ήδη έχουμε, να προετοιμαστούμε ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις υπό Βελγική Προεδρία. Θα είναι πολύ σημαντικό. Συγχρόνως πιστεύω ότι χρειάζεται και μια εκστρατεία ενημέρωσης η οποία έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια το 2009, αυτή πρέπει να ενισχυθεί μέσα στο 2010 πιστεύω. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Τόμσον. Κυρία Ρέντινγκ. Εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, εκτεθειμένες ε, στη βία από τους ε, συντρόφους τους με δραματικές συνέπειες πολλές φορές. Το 2008 παραδείγματος χάνει 157 Γαλλίδες και 65 Ισπανίδες έχασαν τη ζωή τους από άνδρες περισσότεροι από ό,τι έχασαν τη ζωή τους από την τρομοκρατία. Η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε επανειλημμένα στο χάρτη των των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά η βία των ανδρών εις βάρος των γυναικών αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεί αίτιο ανισότητα ε, ανάμεσα στα δύο φύλλα. Σε πρόσφατο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να προτείνει οδηγία για την εξάλληψη κάθε μορφή βία εις βάρος των γυναικών. Και εδώ είναι η ερώτησή μου. Είσαστε ε, πρόθυμοι να αναγνωρίσετε ότι η βία ει βάρο των γυναικών είναι παραβίαση θεμελιωδών θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου προτίθεστε να δρομολογήσετε την εκπόνηση οδηγίας για την απαγόρευση όλων των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών. I absolutely agree with honorable. Συμφωνώ απολύτως. Η βία εις βάρος των γυναικών είναι ένα τρομερό γεγονός και είναι ένα πρόβλημα επίσης το οποίο δεν καταγγέλλεται πάντα. Το 20 με 25% των γυναικών, τουλάχιστον άπαξ διαβίου, υπόκεινται σωματική βία και 10% των Ευρωπαίων γυναικών έχουν υποστεί επίσης και σεξουαλική βία. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει ε, να είμαι πάρα πολύ σύντομη να σας πω τι ακριβώς κάνουμε. Πρώτον πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το οπλοστάσιο των νομικών μέσων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ θα σας κάνω συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών. Ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες όταν συζητάμε τα θέματα της χάρτας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της βίας. Δεύτερον, η συνέργεια η οποία απαιτείται να υπάρχει ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ακριβώς η οδηγία για την, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων ένα πρώτο μέσο αλλά το μέσο αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε και με άλλες δυνατότητες ενισχύοντας σαν παράδειγμα τον ρόλο των ΜΚΙΟ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις στρατηγικές μας ε, ε, για να βοηθήσουμε και την εκπαίδευση των αστυνομικών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να συνεργαστώ με την συνάδελφο Μέλστρομ Έχω την αίσθηση ότι και η χάρτα, όπως επίσης και η δήλωση του Πεκίνου, ε, θα μας βοηθήσουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την διεθνή διάσταση. Εφόσον συμφωνείτε, δώστε μου μία δυνατότητα ε, να πω και ίσως το εξηγήσω αργότερα αυτό, ότι θα ήθελα να υπάρξει επίσης ε, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης καταγγελίας του γυναικείου γενετησίου ακροτηριασμού κάτω από όλες τις μορφές. Είναι κάτι το οποίο έχω ε, στόχο να αντιμετωπίσω άμεσα. Η κυρία Παρβάνοβα, Επίτροπε, ε, πράγματι έχετε εμπειρίες ε, για τις σχέσεις σας με τα μέσα ενημέρωσης και θα προσπαθήσετε να αναλάβετε δράση για να προωθήσετε ε, την αξιοπρέπεια της γυναίκας στα μέσα ενημέρωσης. Να αναφέρω την περίπτωση της κυρίας Άστον, της οποίας οι αρμοδιότητες αμφισβητήθηκαν σε σχέση με τους ε, άλλους τρεις άνδρες οι οποίοι κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ε, θα προστατεύσει την δημοκρασία και την ισότητα στο εσωτερικό των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε στην οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, θα ήθελα όμως να μου πείτε και τι θα κάνετε και με τη στρατηγική δράση σας στο μέλλον ε, και πώς θα βοηθήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί περισσότερο στην επεξεργασία της στρατηγικής αυτής και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ε, νέας στρατηγικής δράσης. Η κυρία Ρέντινγκ. Ο οδικός χάρτης. Ο οδικός χάρτης ισχύει πάντα, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η βία εις βάρος των γυναικών θα πρέπει να είναι ε, κατά προτεραιότητα αντικείμενο αντιμετώπισης. Όλα αυτά θα πρέπει να καταστούν περισσότερο ορατά. Θα υπάρξει μια νέα πολιετή στρατηγική για την ισότητα των ευκαιριών που να βασίζεται ακριβώς στον οδικό χάρτη και ακριβώς μέσω και της, του χάρτη τον οποίο έχει προτείνει ο πρόεδρος Μπαρόσο και ο οποίος δεν πρόκειται φυσικά να αντικαταστήσει την πολιετή μας στρατηγική. Αλλά όλα αυτά θα βοηθήσουν νομίζω και θα επιτρέψουν και στη δική σας Επιτροπή να πάρουν μέρος στις προσπάθειες τις οποίες θα κάνουμε για να συλλάβουμε αυτές τις νέες πολιτικές και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Πώς μπορούμε εμείς να ενισχύσουμε την εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κορνέλισεν. Κύριε Ρέντικ, όπως ξέρετε, αυτή την εποχή εξετάζουμε μία οδηγία για την ε, άδεια τοκετού, προκειμένου να προστατευτεί και η μητέρα και το παιδί. Καταλαβαίνετε ότι επειδή μιλάμε για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι πολύ σημαντική και η άδεια η γονική για τον πατέρα γιατί είναι πάρα πολλοί οι πατέρες οι οποίοι φροντίζουν για το παιδί τους. Ε, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχολούνται και οι δύο οι γονείς. Να κάνουν μπάνιο το παιδί και λοιπά, να το αλλάζουν και λοιπά. Ένα άλλο μέρος του Κοινοβουλίου, οι δημοκράτες κυρίως, πιστεύουν ε, ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική οδηγία για την γονική άδεια για τον πατέρα και να μην συμπεριληφθεί στην ίδια. Οπότε, σας ρωτάω, αν δεν περιληφθεί σε αυτή την οδηγία και η γονική άδεια για τον πατέρα, πιστεύετε ότι θα κάνετε μία άλλη πρόταση προκειμένου να καλυφθούν και οι πατεράδες. Η κυρία Ρέντινγκ. Ναι. Υπάρχει οδηγία για την άδεια τοκετού, όπου η Επιτροπή προτείνει από τις 14 να πάμε στις 18 εβδομάδες. Ήδη αυτή η οδηγία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή για την άδεια τοκετού να περάσει. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να βάλουμε την γονική άδεια για τον πατέρα μέσα σε αυτή την οδηγία. Γιατί φοβάμαι ότι τότε θα χάσει κάθε πιθανότητα να περάσει η οδηγία για την άδεια τοκετού. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ότι είναι ζωτική σημασία και οι πατεράδες να συμμετέχουν περισσότερο στην όλη προβληματική. Και εγώ τρία παιδιά έχω και ξέρω, τρία γόρια Είναι πολύ σημαντικό ο πατέρας να συμμετέχει στην ανατροφή τους από την πιο μικρή ηλικία. Οι κοινωνικοί εταίροι αποφάσισαν για μια γονική άδεια που υποχρεωτικά ένα μήνα παίρνει και ο πατέρας για να μένει στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο λοιπόν, μην το ξεχνάμε. Τώρα όλα τα άλλα, η χονική της ε, η ε, και λοιπά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω πως πρέπει να περάσουν σε μια επόμενη νομοθεσία εφόσον χρειαστεί. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω όλες τις νομικές και όλες τις οικονομικές επιπτώσεις πρώτα απ' όλα. Αλλά θέλω να διαπραγματευτώ όσο γίνεται πιο έντονα με το Συμβούλιο προκειμένου η οδηγία μας για την άδεια το κετού να περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς εμπόδια. Ευχαριστώ. Κυρία Γιανακεδάκη έχει το λόγο. Αναγνωρίζετε ότι το κυρίαρχα κράτη είναι για να καλύτερα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά που αφορούν τους πολίτες τους, ιδιαίτερα σε θέματα εγκληματικής βίας, οικιακή βία, υποχρεωτική γάμη και ε, γενετήσιοι ακροτηριασμοί και πώς θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κυρίαρχα κράτη. Η ερώτηση αυτή βασίζεται στο ότι οι περισσότεροι τομεί στους οποίους αναφέρθηκα είναι θέματα που άπτονται του ποινικού δικαίου στην πρώτη βαθμίδα. Πώς θα υποστηρίξετε λοιπόν τα κυρίαρχα κράτη, κυρία Ρέντινγκ. Προφανώς και θα υποστηρίξουμε τα κυρίαρχα κράτη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σε θέματα ποινικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Το ανέφερα αυτό στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε τις δύο προηγούμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές. επιτροπές συγγνώμη. Στο αστικό πεδίο προχωράμε γρήγορα. Σε ποινικό πεδίο πρέπει να έχουμε πλήρη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και έστω και ένα κράτος μέλος μπορεί να μπλοκάρει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό ακριβώς με τις υπηρεσίες μου, σε συνεργασία με τη Σεσίλια Μέλστρομ, θα εξετάσουμε εκ νέου τις πρωτοβουλίες τις οποίες σκοπεύουμε να αναλάβουμε στον τομέα των ποινικό για να ενισχύσουμε την προστασία των γυναικών. Το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο εντάσσεται στις αρμοδιότητές μου, εμπλέκει τις ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με την στήριξη προς τις γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύματα βίας. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να προχωρήσουμε εύκολα. Να αναφερθώ τώρα στην γενετήσια, στις γενετήσιες ε, μορφές ακροτηριασμού των γυναικών οι συνάδελφοι υπεύθυνοι για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξωτερικές δράσεις και να μην κάνουμε τίποτα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 180.000 γυναίκες στην Ευρώπη κινδυνεύουν να ακροτηριαστούν σε επίπεδο, στο ε, γνωστό επίπεδο και κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα για την πρόληψη ε, του ακροτηριασμού των γυναικών πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει επίσης ε, να ενισχύσουμε και τις έρευνες ε, και την τελική προσπάθεια να την κάνουμε για να μηδενίσουμε το φαινόμενο αυτό στην Ευρώπη. Θα διαβουλευθώ όσο περισσότερο γίνεται με την κοινωνία των πολιτών, θα εξετάσω πολύ προσεκτικά το νομικό πλαίσιο και να νομοθετήσουμε αν χρειαστεί στον τομέα αυτό εφόσον είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε ακριβώς να ορίσουμε και τις κυρώσεις από τη μία αλλά και το τι συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη από την άλλη. Και η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και με την συνάδελφο Σεσίλια Μέλστρομ αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. κυρία Φιγκορέδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε κάποια φάση, κυρία Υποψηφία Επίτροπε, όταν μιλούσαμε για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θυμίζω ότι γιορτάζουμε φέτος 15 χρόνια από την πλατφόρμα του Πεκίνου για τα δίκαια των γυναικών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν ότι απαιτείται να υπάρξει μια χάρτα οι γυναίκες και εξακολουθούν να υφίστανται στην Ευρώπη. Πολλά παραδείγματα δόθηκαν σήμερα, δεν έχω χρόνο να τα επαναλάβω. Είναι λοιπόν βασικό να εμπλέξουμε τις γυναίκες στις διαδικασίες αυτές και αναφέρομαι εδώ στις οργανώσεις των γυναικών, στη συζήτηση η οποία γίνεται. Και γι' αυτό θέτω το εξής ερώτημα. Πώς σκοπεύετε ότι θα πρέπει να εμπλακούν στις διαδικασίες οι οργανώσεις των γυναικών πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών και των οργανώσεών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Η κυρία Ρέντινγκ. Έχω την εντύπωση ότι και στο παρελθόν έχουμε κάνει μια αρκετά καλή δουλειά σε συνεργασία με τις ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα της ισότητας των ευκαιριών στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία αυτή γνωρίζετε ότι το Φόρουμ των Γυναικών, των Ευρωπαίων Γυναικών, θα ε, συνέλθει το Φεβρουάριο για να προετοιμάσει τη συνέχεια της πλατφόρμας του Πεκίνου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν και στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και στη συνάντηση την τελική στη Νέα Υόρκη όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις για τα 15 χρόνια του Πεκίνου. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε έτσι ώστε οι θέσεις μας να γίνουν ε, κατανοητές. Σχετικά με την χάρτα, επαναλαμβάνω ότι γιορτάζουμε την 15η επέτειο της ε, πλατφόρμας του Πεκίνου και ε, έγιναν κάποιες προτάσεις από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα ήθελε να δει να επιβεβαιούνται δημόσια και επίσημα οι αξίες και οι βασικές αρχές των πολιτικών τις οποίες ακολουθούμε. Πολιτικών οι οποίες έχουν πίσω τους μια μακρά ιστορία, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα έχουν και ένα μακρό μέλλον. Γιατί αν μη τι άλλο τα προβλήματα σε πολλούς τομείς παραμένουν. Τα προβλήματα των γυναικών στους χώρους εργασίας, ο συνδυασμός εργασίας και οικογένειας, η συμμετοχή στα επίπεδα λήψης αποφάσεων, Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα υπογραμμίζουν το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Βέβαια μια χάρτα δεν θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα δράσης μας ή τα πολυετή προγράμματα εργασίας τα οποία έχουμε. Μια χάρτα όμως θα επιβεβαιεί προφανώς τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών στα οποία πιστεύουμε. Αυτό είναι το πιστεύω μας και οι αξίες μας. Τελευταία ερώτηση. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σκοπεύετε να εκπονήσετε μια νέα επικοινωνιακή πολιτική που να αφορά αφενός την παρουσίαση στις γυναίκες των πολιτικών μας πέρα από αυτή τη χάρτα που θεωρώ μια θαυμάσια ιδέα αρχών και αξιών, αλλά τις πολιτικές για την καθημερινή ζωή ήταν ένα αίτημα των γυναικών κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών να γνωρίσουν τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο ή η Ένωση για αυτές και από την άλλη πλευρά ε, πώς θα α, εντάξετε τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές της ε, επικοινωνίας στις οποίες ε, θα σχεδιάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέντινγκ. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν αποφάσεις, που θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχετε τις αναλύσεις, έχετε μπροστά σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα καταθέσω εγώ. Γνωρίζετε που ακριβώς ε, βρισκόμαστε ως ε, πρόεδροι μεγάλων επιχειρήσεων. Γνωρίζετε ποιο είναι το ποσοστό μας ε, στα κοινοβούλια, γνωρίζετε όλα τα στοιχεία. Άρα δηλαδή εδώ υπολείπονται πάρα πολλά και η αντιπρόεδρος κυρία Κράτσα έχει απόλυτα δίκιο. Όντως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουμε για να εξηγήσουμε καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε. Και όπως σας έχω ήδη εξηγήσει και προηγουμένως καλή επικοινωνία μπορεί κανείς να έχει μόνο εφόσον έχει και καλή τροφή, καλή ύλη, η ιστορία να είναι καλή. Να ξεκινήσουμε με συγκεκριμένα προβλήματα. Οι γυναίκες στην κοινωνία μας, ε, το τι ε, βιώνουν οι ψηφοφόροι σας και από εκεί να περάσουμε στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ αυτό προτίθεμαι να κάνω στο μέλλον. Νομίζω ότι ε, τα 15 χρόνια από, την, ε, από το συνέδριο του Πεκίνου και ο χάρτης είναι καλά όπλα στα χέρια μας για να προχωρήσουμε. Αργότερα όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Να μην παραμείνουμε στα γενικά ε, ότι δήθεν κάνουμε κάτι για την ισορροπία ανάμεσα δύο φύλλα. Καλό αυτό, αλλά συγκεκριμένα τι γίνεται αν μια γυναίκα θέλει να μείνει σπίτι της, αν θέλει να επανέλθει στη δουλειά, όταν είναι θύμα βίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από συγκεκριμένα παραδείγματα και ε, ας ε, περάσουμε στην πολιτική που ήδη εφαρμόζουμε και πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα στα ε, κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν πράγματι βασίζομαι στους ε, βουλευτές ε, που έχουν την άμεση επαφή με τους εκλογείς τους για να προχωρήσει αυτή η πολιτική επικοινωνίας. Έχουμε άλλα 4-5 χρόνια μπροστά μας μέχρι τις επόμενες εκλογές και θα ήθελα μέχρι τότε όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη να γνωρίζουν τι κάνει η Ευρώπη για αυτές, ε, να ε, γνωρίζουν ε, ποια ακριβώς είναι τα προβλήματά τους και ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει φτάσει η στιγμή για να κλείσουμε αυτό το έντονο απόγευμα. Ευχαριστώ την κυρία Ρέντινγκ ε, που έδειξε τόσο μεγάλη αντοχή. Ευχαριστώ και τις άλλες δύο επιτροπές, ε, την Επιτροπή Γιούρα και τη Λίμπε. Και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών ε, και Ισότητας των Διευθυνών. Ευχαριστώ προφανώς και τις και τους διερμηνείς για τη σκληρή τους δουλειά σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή μας ότι στις 5.30 θα συναντηθούμε στην αίθουσα 1G2. Οι συντονιστές της Επιτροπής ε, θα συναντηθούν εκεί. Και όπως ε, είπα ήδη, ευχαριστώ όλους σας θερμότατα για ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Χαίρετε.